Συνάδελφοι, ας, ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Ας μην καθυστερούμε περαιτέρω. Στην ημερήσια διάταξη έχω λάβει κάποια αιτήματα αλλαγών. Ο κ. Καζά ζητάει το 16 της εσωτερικής αγοράς να αναβληθεί για μια επόμενη συνεδρίαση. Έχει αλλάξει και το χρονοδιάγραμμα και η ψηφοφορία θα γίνει τον Απρίλιο στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Η κυρία Γιάννη Λοβιέτσκαγια σε συμφωνία με τον κύριο Κοστέλο το ζητάει το 19 για την απόσπαση των εργαζομένων και το 38 για τις ε, ενισχύσεις των απόρων να αντιστραφούν σε ό,τι φορά τη σειρά τους. Και το 18 στις το 19. Μετά η κυρία Σαρτιέ, Μωρέν Σαρτιέ, ζητά αύριο να ξεκινήσουμε με την ε, έκθεση πεπραγμένων των τριών τριμερών, των ε, δύο τριμερών διαλόγων. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αν δεν, υπάρχει αντίρρηση, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλάζουμε την μέση διάταξη. Σας ενημερώνω. Ε, ενημερώνω της Προέδρου. Ε, θα χαιρετήσουμε, όχι δεν είναι εδώ, αργότερα. Ε, και δεύτερον ότι η συνεδρίασή μας ε, προβάλλεται μέσω ίντερνετ, μέσω web streaming. Περνάμε στην συζήτηση των νομοδοτήσεων. Έξι σχέδια απαλλαγής ε, ε, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Έχουμε λάβει 15 τροπολογίες εντός των προθεσμιών, 4 για τις τέσσερις ε, υπηρεσίες ε, που εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα ε, για την OFSA 4, για Eurofond 1, 2 για το SEDEFOP ε, και 3 για, το, για την ETF. Και για το συνολικό κείμενο επιδόσεις δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχο των αρισμών λάβαμε μία τροπολογία σε ό,τι αφορά την γενική απαλλαγή για αυτό το κείμενο δηλαδή, την απαλλαγή 2011, λάβαμε τέσσερις τροπολογίες του κύριου Ρή, συμφωνώ με τις τρεις πρώτες, ενώ για την τέταρτη θα έλεγα ότι διαφωνώ με το πρώτο τμήμα. Το συζήτησα και με την Κομισιόν και με την ίδια την υπηρεσία. Σας προτείνω όμως μια προφορική τροπολογία για το δεύτερο τμήμα επαναλαμβάνει την έκκλησή της να διασφαλίσουμε ότι στο φως της εφαρμογής ε, θα πρέπει να αποφευχθεί ε, ε, ε αύξηση των ράλτων, των ποσών που εκκρεμούν προς καθάριση. πέραν του 56% των συνολικών ποσών που είναι διαθέσιμα. Σε ό,τι αφορά το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έλαβα μία τροπολογία του κυρίου Ρή που προτείνει και μια επίκριση ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Μου φαίνεται υπερβολική. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την, ε, για την τροπολογία 2. Έχουμε την τροπολογία 2. Ζητά τα διορθωτικά μέτρα που θα ληφθούν για να διορθωθεί η σημερινή κατάσταση, να ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι είναι μια καλή τροπολογία, καλή Κανένα καλό αίτημα. Προτείνω και μια προφορική τροπολογία που θα επέτρεπε και σε αυτό το κείμενο και στο επόμενο κείμενο να προσθέσουμε την εξής πρόταση. Γι' αυτό το λόγο καλή να γίνει καλύτερη χρήση των, και, των συστάσεων ε, του κέντρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, μεταξύ των οποίων με, μέσα στο πλαίσιο του οποίου και στην ε, ε, κατάρτιση των ε, δικτών και της μακροοικονομικής μελέτης. Σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, προτείνω την, προσω... εξή προσω... Ε, προφορική τροπολογία. Ε, υπογραμμίζει τη συνεισφορά του 2011 του ε, οργάνου αυτού για την επιτυχία των στόχων της Ευρώπης 2020 και ιδιαίτερα για τις ε, πρωτοβουλία πρωτοβουλίας για τη, τα, τις νέες θέσεις εργασίας και δεξιότητες. Ε, καλή την καλύτερη χρήση των συστάσεων της υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την ΟΧΣΑ, σας προτείνω και πάλι μια προφορική τροπολογία προς την ίδια κατεύθυνση. Τα λέγαμε υπογραμμίζει ότι η καλύτερη ε, ασφάλεια και υγεία στο χώρο μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης από το 69% στο 75% που έχει καθοριστεί ως στόχος στην ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020. Και το ίδιο θα το αντικατοπτρίσουμε και στο ε, υπόλοιπο κείμενο, ε, αυτό που σας πρότεινα και προηγουμένως. Τώρα για το ETF. μία προφορική τροπολογία, όχι δύο, τρεις, μία προφορική, στο ίδιο πνεύμα με αυτό που σας παρουσίασα, για την στρατηγική Ευρώπη 2020 που είναι σημαντικό όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα δώσει και δυναμικό για τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες της γειτονίας μας έτσι ώστε να ε, βοηθήσει τις μεταρρυθμιστικές προπάθειες. Γι' αυτό το λόγο έχει σημασία το έργο του ETF στην πρόθεση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Διαβάζει εξαιρετικά γρήγορα η πρόεδρος, δεν γίνεται έτσι. Είναι η ίδια παρόμοια τροπολογία με αυτή που σας είχα πει προηγουμένως. Μιλάμε ε, για την καλύτερη χρήση των συστάσεων κλπ. κλπ. δύο άλλες τροπολογίες από τον κύριο Ρήμια που λέει, υπενθυμίζει ότι ε, το θέμα του Ιταλικού, το Ιταλικό θέμα το οποίο δεν είναι ακόμα, παρόλο ότι η Κομισιόν ζήτησε να ε, έχει στηθεί από την Κομισιόν λύσει το πρόβλημα, ε, είναι το θέμα του ε, τοπικού προσωπικού και ο κ. Συρκά έχει υποβάλει μια τροπολογία. Δεν χρειάζεται προσωπική τροπολογία γιατί το πρόβλημα τους, της σύμβασης δεν είναι πρόβλημα σχετικό με την Κομισιόν, δεν αφορά την Κομισιόν, αλλά τη χώρα και τις περιφερειακές αρχές. Γι' αυτό το λόγο θα υποβάλω μια προφορική τροπολογία για να διευκρινίσω αυτή την πρόταση. Και μετά υπάρχει και μια τρίτη τροπολογία της κυρίας Αρκίν, την οποία μπορώ να δεχτώ που αναφέρεται στις δεσμεύσεις της υπηρεσίας αυτής για την καλύτερη χρήση, για την καλύτερη διαχείριση των δαπανών της. Και τέλος για την υπηρεσία για την κατάρτιση, όχι, όχι, για το συνολικό κείμενο, το οριζόντιο κείμενο για την απαλλαγή 2011, επιδόσεις δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχο των οργανισμών, Έχουμε μια τροπολογία του Jean Lambert που προτείνει να διοργανωθεί καλύτερα η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών αρχών. Σας προτείνω να δεχτούμε αυτή την τροπολογία και να προσθέσουμε και μια προφορική τροπολογία που θα αναφέρεται στην βασική μας ανησυχία την οποία σας ανέφερα στα προηγούμενα κείμενα. Σας προτείνω να ανοίξουμε τη γενική συζήτηση, ο κ. Σωρή. Ευχαριστώ. Δεν έχω και πολλά να πω. Σημειώνω το γεγονός ότι οι περισσότερες τοπολογίες έχουν γίνει δεκτές από την εισηγήτρια. Θα δούμε τι θα γίνει με την ψηφοφορία. Εγώ τις υποστηρίζω. Υποστηρίζω όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Α, θέλει καλή άλλο το λόγο. Ο κύριος Σέρκας. Η ομάδα μας, Πρόεδρε, συμφωνεί απόλυτα με τις τροπολογίες οποίες αναφέρατε ή διαβάσατε. Και μία ακόμα φορά θα υποστηρίξουμε με αυτόν τον τρόπο το έργο των υπηρεσιών αυτών, των οργανισμών αυτών, που μα βοηθούν τόσο πολύ να πετύχουμε του στόχου τη στρατηγικής Ευρώπη 2020 και, να, βγούμε από την κρίση. από πλευρά τη ομάδα μας, υποστηρίζουμε τις τροπολογίες έτσι. Ευχαριστώ. Κομισιόν θα ήθελε το λόγο. Όχι. Είναι συμφωνή. Τα τρία μηνύματα τα οποία εγώ συγκρατώ για αυτό το δίκτυο, για αυτό το πακέτο, είναι πρώτον η απόλυτη ανάγκη να βελτιστοποιήσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και τις, ε, και τις υπηρεσίες αυτές, ε, που μεταξύ αυτών έχουμε και τέσσερις που εμείς στη δική μας αρμοδιότητα, που είναι εξαιρετικά καλές, ε, πολύ αξιόλογες, μετά έχουμε την υπηρεσία του, ε, του Τωρίνου και την ε, σύμβαση εγκατάστασης. Δεν βρίσκω τη λέξη στα γαλλικά. Α, τη συμφωνία ε, για τον καθοσμό της έδρας. Παρακτοξώ γιατί συνήθως οι τοπικές αρχές τρελαίνονται να φιλοξενούν τέτοιου είδους υπηρεσίες και να τις διευκολύνουν. Τώρα δυσκολευόμαστε με τις τοπικές αρχές, τέλος πάντων παράδοξο λίγο. Είναι πρόβλημα επικουρικότητας, από ό,τι καταλαβαίνω είναι θέμα εθνικών και περιφερειακών, υπερφερειακών και τοπικών αρχών. Η δική μου ανησυχία επιπλέον αφορά το ΣΕΝΤΕΦΟΠ απουσία διευθυντή εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση, αλλά δεν είμαστε και οι μόνοι που κάνουν αυτή την παρατήρηση. Σημείο 9. Ο κ. Μπλόγο είναι εδώ ή έχει αντεκατασταθεί. Έχει έκθεση. Δεν ξέρω σε ποια συνεδρία είναι αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να είναι εδώ ε, ο κ. Μπουλόν. Θα μπορούσαμε να περάσουμε στο 10 ενδεχομένω. Ε, έκθεση Steinruck. Οι σκιώσεις ηγητές είναι εδώ. Ο κ. Σωρή, ο κ. Μπενιό είναι εδώ. Η κυρία Λομπέρ και η κυρία Τσούμπερβεν. Θα έρθει σύντομα. Λοιπόν, περνάμε στην έκθεση Steinruck. Εφαρμογή τη οδηγία 2004-25 σχετικά με τι δημόσιε προσφορέ εξ αγοράς. Θα εξετάσουμε τις ε, τροπο, τροπολογίες, 7 συγκεκριμένα. Ε, τη βάση τροπολογιών που είχαν κατατεθεί Πρόκειται για γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Γιούρη. Ε, εξηγητής εκεί είναι ο κ. Λίνο, ο πρόεδρος της Επιτροπής δηλαδή. Ο κ. Στάινρουκ έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Εν ώψη της προ... προηγούμενης συζήτησης όλοι υποθέσαμε ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Αλλά το ότι οι ομάδες ε, θα μπορούν να συνεργαστούν μετά από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν ε, καταφέραμε μόνο με μία συνάντηση να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους για αυτό το έξοχο πνεύμα συνεργασίας και έτσι επιτύχαμε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την πλευρά των εργαζομένων και την αρχή της συναπόφασης και από την άλλη να διατηρήσουμε την, το ενδιαφέρον και τις δραστηριότητες της, του οικονομικού τομέα. Ως ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες ήταν πάρα πολύ ε, σημαντική για μας η κάλυψη της πτυχής των εργαζομένων έτσι ώστε όταν υπάρχουν αναδιαθρώσεις ή συγχωνεύσεις ή μεταβιβάσεις να έχουν και αυτοί το λόγο, να ακούγεται η φωνή τους, να ενημερώνονται και να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα με το συμβιβασμό. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν δείξει πνεύμα συνεργασίας και όλα βαίνουν καλώς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα όσα ακούσαμε από την κυρία Στάινμπρουκ. Στην αρχή φοβόμασταν λιγάκι, γιατί θεωρούσαμε ότι ίσως όλα αυτά δεν είναι τόσο ρεαλιστικά. Καλές προθέσεις δηλαδή για τους εργαζόμενους αλλά ίσως σκεφτήκαμε ότι είναι λίγο υπερβολικά. Εν πάση περιπτώσει, μετά από διαπραγματεύσει συμφωνήσαμε και έχουμε φτάσει και σε συμβιβασμού. Αυτοί οι συμβιβασμοί λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων, χωρί ε, μπλοκαρίσματα, χωρί τροχοπέδε στη συνήθη λειτουργία των επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν συμβιβαστικέ αυτέ τροπολογίε, τι οποίε μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ο Φιλιμπένιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το επικοδομητικό πνεύμα στην συνάντηση των σκιωδών και τις πολύ θετικές προτάσεις για συμβασμούς. Είχαμε κάποιες θεμελιώδεις ε, διαφορές βέβαια, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι κάτι που μπορούμε γενικά να το υποστηρίξουμε. Στη συνάντηση των σκιωδών συμφώνησα να υποστηρίξω όλες τις συμβαστικές τροπολογίες εκτός από μία, έξι δηλαδή από τις 7 υπήρχαν πολλές παραχωρήσεις που έγιναν από πολλές πλευρές τελικά και νομίζω το κείμενο, το κείμενο ήταν γενικά αποδεκτό. Δεν θα υποστηρίξω όμως την συμβαστική Α ως έχει, γιατί δεν θεωρώ ότι το να αντιταχθούμε σε περαιτέρω, απελευθέρωση ή απορρίθμιση, εν και η ιδέα ότι η απελευθέρωση είναι κάτι αρνητικό, δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο βέβαια. Και οποιασδήποτε μελλοντικέ αλλαγέ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να είναι κατάλληλε. Παρά να πούμε ότι δεν είμαστε υπέρ μια περαιτέρω απελευθέρωση. Αυτή είναι μια μικρή όμω επιφύλαξη. Είμαι ικανοποιημένο γενικά από τη δουλειά που έγινε, από την ε, στάση τη ε, εισηγήτρια και από τη στάση των συναδέλφων από τι άλλε ομάδε. Θέλει κανένα άλλο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εδώ, ούτως ή άλλως. Θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Μια σύντομη παρατήρηση μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφός μου οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης που έχει γίνει μέχρι τώρα πρέπει να τις μελετήσουμε, να τις αναλύσουμε διότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και για τις δύο πλευρές και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους και βεβαίως μας, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι επιπτώσεις για τους εργαζόμενους όμως τα τελευταίες δεκαετίες μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ε, απελευθέρωσης, φιλελευθεροποίησης της, ε, του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που να μην είχε αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Καμία. Γι' αυτό ακριβώς το θέσαμε έτσι. Ωραία. Εν τη αυτή περίπτωση, μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο για την εκνομοδότηση αυτή και η νομική υπηρεσία θα αποφανθεί στις 19 Μαρτίου. Η εισηγήτριά μας ε, έχει την αμέριστη εμπιστοσύνη μας, ούτως ώστε να μας υποστηρίξει στο εσωτερικό της, νομικής, της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα επίσης ε, σε όλους να παρακολουθήσετε τι ε, τις διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων όταν λάβουν χώρα αυτές τις διαπραγματεύσεις και στη συνάντηση των σκιωδών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα περάσουμε τις απόψεις μας και γενικά μπορούμε να τις περάσουμε όταν θέλουμε να, να υιοθετηθεί κάποια γνωμοδότηση. Ο κύριος Μπουλό είναι εδώ. Όχι, δεν θα μιλήσω ο βοηθός του. Πρέπει να περιμένει τώρα όλη η Επιτροπή. Είναι 9.30. Υποτίθεται ότι θα το συζητούσαμε 9 και 20 αυτό το σημείο. Η κυρία Μωρίς Σαχτιέ, η κυρία Χίρσα. Η κυρία Σαχτιέ θέλει να μας μιλήσει για το τι διαμήθη στον ε, τριμερή διάλογο για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Βεβαίως. Μια στιγμή, μια στιγμή. Μια στιγμή. Για να τα πω λίγο επίσημα τα πράγματα, έτσι, για το web streaming. Λοιπόν, ε, επιταχύναμε λιγάκι τις εργασίες μας και θα πάμε στο σημείο 41. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τι ε, διαπραγματεύσει ε, στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο για την οδηγία που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έχετε το λόγο κύριε Συγήτρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους εδώ της Επιτροπής Απασχόλησης για την εξέλιξη αυτού του τριμέρου διαλόγου ε, μετά από μια πρώτη συνεδρίαση επαφών μέσα στον Ιανουάριο, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία ακριβώς, όπου διαισθανόμαστε ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες λόγω του ότι έπρεπε το Συμβούλιο να μπει στην ουσία του προβλήματος και σε όλα τα προβλήματα που θέτει αυτή η νέα οδηγία λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι εξόχως τεχνική. Κάναμε λοιπόν την πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του ε, διαλόγου χθες το βράδυ και σε αυτή την πρώτη συνάντηση ξεχερσώσαμε έτσι το έδαφος, ε, συζητήσαμε διάφορα σημαντικά σημεία τα οποία, στα οποία δεν υπάρχουν διαφωνίες. Στην Επιτροπή Απασχόληση έχουμε μια μέθοδο εργασίας και αυτή ακριβώς επικυρώθηκε. Ε, γιατί θέλαμε το κείμενό μας να πλησιάσει στο κείμενο του Συμβουλίου, το οποίο από προεδρία σε προεδρία είχε εξελιχθεί πάρα πολύ και εμεί με τις τροπολογίες μας θέλαμε να πλησιάσουμε αυτή τη θέση του Συμβουλίου. Ε, καθώς αλλάζουν Προεδρίε, εμείς, βλέπαμε διαφορετικέ θέσει μπροστά μας και δυσκολευόμαστε εξαιτία αυτού. Χάρη στη δουλειά που κάναμε εδώ στην Επιτροπή Απασχόληση ε, φτάσαμε σε πολλά σημεία ε, τα οποία τα συμφωνήσαμε. Ποια είναι τα υπολείμματα τα οποία ακόμα συζητάμε. Πρώτον, μέτρα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Το Συμβούλιο ήρθε με έναν εμπειρογνώμονα. Και ευτυχώς, χάρη στην ομάδα εργασίας και στη δουλειά που είχε κάνει, ε, ο εμπειρογνώμονας είχε δώσει τις απόψεις του και άρα κερδίσαμε κάποιο χρόνο. Έπρεπε λοιπόν να συμφωνήσουμε για μια διατύπωση των ε, μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και της επαγρύπνησης που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αν υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά, εν τη αυτή περιπτώσει θα έχουμε μια ευρωπαϊκή αντίδραση άμεση, χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο σημείο είναι η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας. Θα θυμάστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο διαρκεί τώρα χρόνια θα πρέπει να βγούμε από αυτό το άδεια έξοδο. Ε, το 2004 φτάσαμε σε μια οδηγία που ήταν ανεφάρμοστη. Και χθες το βράδυ η πρόταση του Συμβουλίου και της Κομισιόν ήταν να έχουμε μία τριετία για την μεταφορά αυτής της οδηγίας. Δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά η θέση μας ήταν και, είχαμε, και συμφωνούσαμε με τους κοιόδης εισηγητές είναι να ζητήσουμε μια συρρήκνωση της προθεσμίας από τρία χρόνια σε δύο χρόνια γιατί είναι μια ιστορία που κρατάει αρκετούς μήνες και έχουμε μια οδηγία που δεν εφαρμόζεται από το 2004 ούτως ή άλλως ε, την προθεσμία που θα θυμάστε μέσα στην οποία θα μπορούμε να εργαστούμε μέχρι τον Νοέμβριο, όχι Οκτώβριο 2013, ενώ θέλουν να μας επιβάλλουν ε, προθεσμία μέχρι τον Απρίλιο του 2014 και αυτό ήταν στη λύση, γιατί ακριβώς πέφταμε πάνω στις ε, εκλογέ και θα ήταν αυτό ένα πολύ κακό μήνυμα που θα δίναμε για την εξέλιξη αυτού του φακέλου. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μία ε, προθεσμία διετίας για τη μεταφορά αυτής της οδηγίας σε εθνικές νομοθεσίες. Αυτό προκάλεσε μια έκπληξη. Δεν είναι ο συνήθις ρυθμός εργασίας. Παράλληλα θα πρέπει να εκπονήσουμε και τον πρακτικό οδηγό, που είναι πολύ χρήσιμος. Ε, θέλουμε να υπάρχει μια σχέση όμως ανάμεσα στον πρακτικό οδηγό και στην εφαρμογή της οδηγίας, τη μεταφορά της οδηγίας. Γιατί αν έχουμε τον ε, πρακτικό οδηγό ε, έτοιμο μετά τη μεταφορά δεν έχει νόημα. Ζητήσαμε λοιπόν στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα γίνει στις 26 Μαρτίου να υπάρχει ένα σχέδιο εργασίας ε, της Κομισιόν και για τον πρακτικό οδηγό αυτό και κάποιες προβλέψεις για την προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας. Αυτά πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Στο μεταξύ ελπίζω να έχει φτάσει και ο εισηγητής που περιμένετε. Αυτά κάναμε χθε το βράδυ με εσά και με το σύνολο των σκιωδών εισηγητών. Και χρήσιμο θα ήταν να ακούσουμε την άποψη της Κομισιόν για αυτή την διετία, που... την προθεσμία ας πούμε, της διετίας. Προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια τάση προς την συρρήκνωση της προθεσμίας. Ο κ. Σέρκας. Η συγγήτριά μας, η κυρία Ράπτη, προσπάθησε να φτάσει, αλλά εξαιτία της αλλαγής ε, της ημερησίας διάταξης δεν τα έχει καταφέρει. Ε, μου είπε όμως να σας ενημερώσω για τρία πράγματα. Καταρχήν, όπως είπε η κυρία Μωράν Σάρτιε, η συνάντηση ήταν πολύ θετική, πολύ επικοδομητική. Οι προτάσεις μας είναι κοινέ. η κυρία Ράπτη είναι πολύ ικανοποιημένη και ελπίζει ότι έτσι θα συνεχιστεί και μέχρι τέλος όπως η κυρία Μωρά, ε, ε, μένουν, τα δύο, μένουν δύο αυτές εκκρεμότητες, τις ε, οποίες καλό είναι να τις ε, ε, πολεμήσουμε μέχρι τέλους. θα πρέπει να δούμε αν θα αλλάξουν τα επιστημονικά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πιέσουμε και την Κομισιόν, η οποία είχε ήδη 8 χρόνια στη διάθεσή τη για να κάνει όλε τι μελέτε που χρειαζόντουσαν, για να μην ε, χρειαστούν τρία χρόνια ακόμα για να μεταγραφεί η οδηγία, που έτσι κι αλλιώ ε, ε, δεν πρόκειται για την βίβλο στις παλαιότερες και νεότερες εκδόσεις της. Ας σπρώξουμε λίγο τα πράγματα, να τρέξουν πιο γρήγορα για να κλείσει το θέμα. Ε, αν δώσετε το λόγο στην ε, Κομισιόν θα ήθελα να ξέρει η Κομισιόν ότι οι δύο βασικές ομάδες, οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ε, της Ευρωβουλής ε, συμφωνούν να δοθεί μια όθηση. Υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτές που θα θέλαν το λόγο. Ο κ. Κλάρκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξετάζοντας τις τροπολογίες, εν συντομία, ε, αναφέρονται στην έκθεση του οφθαλμού και στη δόση αυτή, στο όριο σε δύναμης δόσης και λέει ότι πρέπει να είναι 50 MSV ανά έτος. Η τροπολογία 8 λέει ότι πρέπει να είναι 50 και η 7 λέει πάλι 50 και η 38 λέει 15 μιλισίβερ το χρόνο για τον φακό των οφθαλμών. Δεν ξέρουμε τελικά πόσα MSV ε, προτείνονται. Η πρόεδρος, δεν νομίζω να μιλάτε, εμείς μιλάμε για το 40, για το 15 λέει ο κ. Κλάρκ δεν μιλάμε. Όχι, όχι, είμαστε σε άλλο θέμα λέει η πρόεδρος διότι η δεν ήταν εδώ, δεν είναι εδώ και είμαστε στο 41 41 ηλεκτρομαγνητικά πεδία Αχ, ζητώ συγγνώμη λέει ο κύριος Κλάκ. δεν πειράζει λέει η πρόεδρος λοιπόν η Κομισιόν Πέρα από αυτά που ακούσαμε για τα όσα δημιούργησαν χθε στον τριμερή διάλογο, θα ήθελε να παρέμβει και να μας πει, να μας διαβεβαιώσει ότι υπάρχει καλή θέληση από πλευρά της για την εφαρμογή της οδηγίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η θέση της Κομισιόν, παρότι δεν είχαμε προβλέψει να πάρουμε το, το λόγο σήμερα εδώ, την εκφράστηκε χθε στον τριμερή διάλογο. Επαναλαμβάνω απλώ ότι θα λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το γεγονός ότι οι δύο μας θέλαν να, προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Η δική μας άποψη είναι ότι η οδηγία όντω υιοθετήθηκε με καθυστέρηση, όντω υπήρξαν πολλέ συζητήσει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Παρ' όλα αυτά, ε, αν χρειαζόμαστε τρία χρόνια για να την εφαρμόσουμε σωστά, χρειάζονται τρία χρόνια. Τέρμα. Τέλο πάντων, παρ' όλα αυτά, θα λάβουμε υπόψη τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο των ε, διαπραγματεύσεων, απλώ εδώ εκφράζω τη θέση όπω εκφράστηκε και χθε το βράδυ. Κύριε Σαχτιέ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και ευχαριστώ όλους όσους ε, εργάστηκαν επί του θέματος και μας υποστηρίζουν. Το μόνο που θέλω να πω είναι, και να υπενθυμίσω στους συναδέλφους, είναι ότι όλος ο χρόνος που κερδίζουμε για το φάκελο αυτό, το κερδίσαμε χάρη στο Κοινοβούλιο, χάρη σε μια πιο αποτελεσματική μέθοδο εργασία, γιατί δεν είμαστε εμείς που καθυστερήσαμε τις διαδικασίες. Επομένως, έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε απαιτητικοί για... και να απαιτήσουμε έτσι μια επιτάχυνση και από τους εταίρους μας. Νομίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης ζητούν το ίδιο. Θέλουμε ε, μεταφορά σε δύο χρόνια, όπως αρχικά είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό θέμα. Γνωρίζω λιγάκι περί πρόκειται. Ε, αλλά και επειδή ακριβώ το γνωρίζω λίγο περί τίνο πρόκειται, ξέρω ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη. Στι 26 Μαρτίου θα γίνει ο επόμενο τρίλογο και μέχρι τότε θα έχουμε λάβει τι ε, απόψει τη Κομισιόν και του Συμβουλίου, τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό στον δεύτερο αυτόν επίσημο τριμερό, τριμερή διάλογο. Πάμε τώρα στο σημείο 9, επιτέλου τη ημερησία διάταξη. Ο κ. Μπουλό είναι μαζί μα και μπορούμε να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Ανάπτυξης σχετικά με την δημιουργία ενός σώματος ενό Ευρωπαϊκού Σώματο Εθελοντών Ανθρωπιστική Βοήθεια. Υπάρχουν πέντε συμβαστικέ τροπολογίε που κατατέθηκαν μετά από τι 44 τροπολογίε που είχαν καταθέσει διάφοροι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Μιλούσα ε, για τα θέματα, ε, ε, τα προβλήματα μάλλον της ιατρικής δημογραφίας ε, στη Ρουμανία. Λοιπόν, Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σώμα ατόμων που παρεμβαίνουν σε χώρους όπου έχουν συμβεί καταστροφές ε, για ανθρωπιστικούς λόγους, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτύξει τη δράση της η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο γρήγορα, πέρα από αυτά που κάνει ήδη. Έχω 69 τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην σύνταξη αυτής της έκθεσης και των συμβασμών. Ε, των, ε, και των σοσιαλιστών και των πράσινων και των φιλελεύθερων που μας επέτρεψαν να ομαδοποιήσουμε σε πέντε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και σε μία προφορική. Σε αυτές, σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες δημιουργήθηκαν συνενέσεις για την επιλογή και την, και την κατάρτιση των ατόμων που θα πρέπει να βρούμε, ούτω ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις. Και μέσα από αυτές τις τροπολογίες ε, λέμε ότι η κατάρτιση θα πρέπει να είναι ποιοτική και ότι το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας ανάμεσα στους εθελοντές και του οργανισμού που τους στέλνει στον τόπο της καταστροφής θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ε, ούτως ώστε να ξέρουν οι μεν και οι δε υποχρεώσεις. Επίσης, οι επιλεγόμενοι εθελοντές θα πρέπει να έχουν μια συνεχή κατάρτιση, ούτως ώστε η εμπειρία που αποκτούν μέσα από την παραμονή τους στους τόπους αυτούς να θεωρείται ως μαθητεία που θα τους επιτρέψει εν συνεχεία να ζητήσουν και να βρουν μια νέα θέση. Η βασική ιδέα που προκύπτει από αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και εδώ ευχαριστώ ακόμα μια φορά τους συναδέλφους ε, και είμαι στην ε, διάθεσή τους μπορώ λοιπόν να σας πω ότι μπορώ να απαντήσω κάλλιστα σε όλες τις παρατηρήσεις σας. Η κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, μπορούμε να υποστηρίξουμε όλες τις τροπολογίες και τις ιδέες ε, του κυρίου Μπολάν. Μπουλάν, υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία τονίζουν την σημασία της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των εθελοντών επίσης ε, ε, την κάλυψη του κόστους ασφάλειας και προστασίας και πιστεύουμε ότι έχουμε καταλήξει σε έναν πολύ καλό συμβιβασμό και θα συστήσω στους συναδέλφους μου να υπερψηφίσουν αυτέ, αυτούς τους συμβιβασμούς και τις, ε, ε, τις τροπολογίες και τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Κυρία Χάρκιν. I too would like to thank the rapporteur for... Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία. Καταλήξαμε σε πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες εξετάζοντας αυτή τη γνωμοδότηση. Γνωρίζαμε ασφαλώς τις συνθήκες των εθελοντών και σε τι συνθήκες και καταστάσεις εργάζονται και σε τι, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν και κινδύνους και εξετάσαμε τι μπορούμε να, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κοινωνική ασφάλιση. Παραδείγματο χάρη, και πιστεύω ότι υπάρχουν τροπολογίες που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Επίσης συμπεριλάβαμε σε ένα συμβιβασμό, σε μία συμβασική τροπολογία, το γεγονός ότι οι εθελοντές πρέπει, πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία αν θέλουν να, να αναλάβουν ένα ρόλο μαθητευόμενο, μαθητευόμενο ε, άρα λοιπόν πρέπει να προσφέρουμε και αυτές τις ε, ευκολίες κατάρτισης ε, εφόσον το επιθυμούν. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και θα υπερψηφίσουμε και εμείς. Ευχαριστώ. Ζητά κανείς άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Κύριε Μπουλόν, χρειάζεται ξανά το λόγο. Όχι, ε. Τέλεια. Θα ψηφιστεί αύριο. Περνάμε στο σημείο 11 της ημερησίας διάταξης. Δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Χίρς. Θα μας παρουσιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. γνωμοδότηση υπόψη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. της οποίας εισηγητής είναι ο κύριος Άλμπρεχτ. Κυρία Χίρς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας δώσω μία σύντομη επισκόπηση των ε, τροπολογιών τις οποίες έχουμε επεξεργαστεί. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές. Είχαμε τρία, τρεις συναντήσεις ε, μέχρι τώρα και επιτύχαμε πάρα πολύ να συγκεράσουμε αντίθετες και αντιμαχόμενες απόψεις. Πιστεύω ότι έχουμε συμφωνήσει ε, γενικά στις γενικές γραμμές και αύριο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε τρεις συμβασικές. Ε, η πρώτη αναφέρεται σε αυτό το, την μαύρη λίστα, blacklist, όπου ο στόχος είναι να απαγορεύσουμε ε, στους εργαζόμενους που είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και να μπουν στην, ε, στη μαύρη λίστα και να υποστούν διακρίσεις, αρνητικές διακρίσεις και γενικά αρνητική μεταχείριση. Εδώ συμφωνήσαμε όλοι. Το δεύτερο σημείο, σημείο στο οποίο δεν έχουμε απολύτως καταλήξει είναι η έγκριση ε, μεταξύ ε, εργαζομένων και εργοδοτών και η συμφωνία δηλαδή ε, που πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να δώσει την έγκρισή του, την άδεια δηλαδή, για τον χειρισμό των προσωπικών του δεδομένων, όποτε το ζητήσει η εργοδοσία. Ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα δεδομένα ενός εργαζόμενου όπως τα παιδιά που έχει, που πηγαίνουν σε ποιο παιδικό σταθμό, ε, προσωπικά στοιχεία. Γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς η έγκρισή του. Τώρα η συμβιβαστική 10 ε, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Το SEED, ο επόμενος συμβιβασμός αναφέρεται ότι εφόσον ζητείται η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα πρέπει να έχει ε, πλεονεκτικές επιπτώσεις ε, στον εργαζόμενο ε, και θα πρέπει επίσης για τους εργαζόμενους να υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα. Παρεμβάλαμε και έναν άλλο συμβιβασμό, το G1, που λέει, συμβαστική τοπολογία δηλαδή, που λέει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει στην όλη διαδικασία. Να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία. Συνεχή έχουμε τις συμβαστικές ε ε και F εδώ είχαμε, ακούσαμε διάφορες προστάσεις για τον αριθμό, η δηλαδή μεταχείριση και επεξεργασία των δεδομένων. 250, ε, 250 είπαμε ότι μπορούν ε, περιπτώσεις να ε, υποστούν επεξεργασία κατόπιν ετήσως και εν συνεχεία είχαμε την ε, συμβιβαστική τροπολογία που βασίζεται στο άρθρο 82 η οποία λέει ότι θα πρέπει άρθρο 82 λογική σκέψη 124 που λέει ότι εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την επεξεργασία δεδομένων ε, θα πρέπει να γίνει πρώτη αναφορά στο, στην αιτιολογική σκέψη 124. Αυτό υπάρχει στην τροπο, ε, συμβαστική G. Στο H, ήτα, λέμε ότι θα πρέπει, αν υπάρχει ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτη χώρα, να εφαρμοστούν οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 ε, τρο, συμβιβαστική ε, I, συγγνώμη, γιώτα. Εδώ πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές και έχουμε βάσει του άρθρο 86 ε, θέλουμε να ληφθούν, να ληφθούν υπόψη και οι δαπάνε. Το κόστος ε, δηλαδή όλες τις ε, διαδικασίες επεξεργασίας, διότι αυτό έχει επιπτώσει στις μικρές επιχειρήσεις. Στο, στη συμβαστική J, J εδώ θέλουμε να εισαγάγουμε μια σχετική ευελιξία των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού δεδομένου ότι οι βασικές αρμοδιότητες ανήκουν στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών αλλά θέλουμε να εισαγάγουμε και το στοιχείο της ευελιξίας. Ξέρω ότι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πέραν του ενός ε, κρατών μελών ε, θέλουν να καλυφθούν νομικά για όλες αυτές τις διαδικασίες δεδομένων. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό το στοιχείο της ευελιξίας. Και τέλος θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων να γίνονται ε, ιδίως από δεσπόζουσες εταιρείε μέσα στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής. Τώρα πιστεύω πιστεύω ότι έχουμε διευκρινίσει και διάφορα, διάφορες παρανοήσεις που έγιναν αρχικά λόγω μεταφράσεων, αλλά πιστεύω το κείμενο τώρα είναι σωστό, οι μεταφράσεις είναι ακριβείς. Η... Επίσης δεν θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα αποφυγής ή παράκαμψης του κανονισμού σε περιπτώσεις που υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Να μην ε, παρουσιαστεί αυτό ως δικαιολογία παράκαμψης ή παρέκκλησης. Παραδείγματο χάρη, εάν μία εταιρεία ε, επιτρέπει, ε, επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων μπορεί να γίνει μία... Α, ε, την χρήση κινητών τηλεφώνων ε, και την κατακράτηση στοιχείων, έτσι. Εάν λοιπόν επιτρέπει τη χρήση κινητών και τη καταγραφή των δεδομένων και αν χαθεί το κινητό τηλέφωνο, τότε θα πρέπει να σβηστούν και όλα τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να υπάρχει μία, ένας διαχωρισμός ε, μεταξύ του αν υπάρχει εταιρική συμφωνία ή συλλογική σύμβαση. Και αυτά αναφέρονται ή στο ένα ή στη μία ή στην άλλη συμφωνία, στο πλαίσιο. Και ε, ο συμβιβαστική ΚΑΠΑ, K, αναφέρεται στα ελάχιστα πρότυπα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να πρέπει να ενημερώνονται ε, ότι γίνεται κάποια, διαπραγμα... κάποια παρακολούθηση έτσι ώστε να αποφύγουμε πάση θυσία οπτικοακουστικές παρακολουθήσεις και θα πρέπει να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι ε, σε τέτοια περίπτωση αν παρακολουθούνται ή γιατί, για ποιο λόγο να είναι όλα διαφανή. Αυτό το οποίο ακόμα κρεμεί είναι κατά πόσον μπορούν δεδομένα να χρησιμοποιηθούν για προληπτικούς λόγους υγείας. Αυτό δεν το έχουμε λύσει. Παραδείγματος, ναι, παραδείγματος χάρη δεδομένα υγείας που αφορούν τους εργαζόμενους και επίσης η, το θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα emails ε, πώς θα γίνει η διαχείριση αυτών των δεδομένων. Αυτά είχαμε συζητήσει επίσης τις πράξεις εξουσιοδότηση και την χρήση τους. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό να τα συζητήσουμε, αλλά στην Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων εξετάζονται λεπτομερώς οι πράξεις εξουσιοδότηση από τις διάφορες ομάδες και γι' αυτό η δουλειά αυτή γίνεται ήδη, αλλά δεν χρειάζεται να ε, επαναλάβουμε όλη αυτή την εργασία. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους συνεργάτες για την εξαιρετική εργασία που, που έκαναν. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη ε, συμβιβαστική λύση. Δεν θα είναι τέλεια, αλλά θα είναι η βέλτιστη. Ευχαριστώ. Κυρία Λάμπερτ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Um, και ευχαριστούμε πραγματικά την, τον ε, εισηγητή, ήταν, την εισηγήτρια, ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία μας και βεβαίως μπορούμε να υποστηρίξουμε την πλειοψηφία ε, των συμβαστικών τροπολογιών συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας, της K. Διότι υπάρχουν και θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας που εμπλέκονται εδώ πάντοτε στα δεδομένα. Υπάρχουν ακόμα μερικά προβλήματα όπως ανέφερε και η συγγήτρια. Ένα το μέσο με δυσκολεύει είναι ο βαθμός της ευελιξίας που θα πρέπει να δοθεί στις ε, συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων και εάν αυτές οι συμφωνίες πρέπει να τηρούν το επίπεδο του κανονισμού ή εάν θα επιτρέπεται κάποια παρέκκληση από αυτά τα πρότυπα. Ε, το θέμα είναι να μην μειώσουν τον πύχη ε, του, επίπεδου, του βασικού επίπεδου που ορίζει ο κανονισμός εμείς δεν θέλουμε διόλου οι συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων να υποσκάπτουν τον κανονισμό και να χαμηλώνουν τον, τον πύχη της ουσίας του κανονισμού. Ε, γι' αυτό έχουμε και ορισμένες επιφυλάξεις στη συμβαστική τροπολογία J. Αν και τα περισσότερα τα υποστηρίζουμε στην συμβαστική J, αλλά έχουμε ακόμα επιφυλάξεις. Τώρα, όσον αφορά ε, αυτά που ελέγχθησαν για τις πράξεις κάτι εξουσιοδότηση. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια και πιστεύουμε ότι η, πρα... η Επιτροπή θα έχει μια γενική εικόνα του κανονισμού και θα ξέρει ακριβώς πότε χρειάζονται και πότε δεν χρειάζονται. Δεν λέω ότι είμαστε ερωτευμένοι και ένσερμοι υποστηρικτέ των πράξεων κατεξουσιοδότηση εξουσιοδότηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται και να διαγραφούν τελείω. Εν πάση περιπτώσει εμείς πιστεύουμε ότι ε, αυτή η συζήτηση για τις πράξεις κάτι εξουσιοδότηση πρέπει να γίνει όταν θα έχουμε μια γενική εικόνα του τι προτείνει ο κανονισμός στο σύνολό του. Ε, ζητάει κανεί το λόγο τον κύριο Σέρκα. Ο κύριο Γκορεάνο πριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Χίρς και τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές. Ήταν μια έντονη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Φτάσαμε νομίζω σε καλές συμβαστικές τροπολογίες. Και σε ό,τι αφορά το ΕΛΚ, ε, εμείς ε, τις υποστηρίζουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Καμία διαφωνία με τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Αλεχάνδρο Θέρκας. Και εμείς θέλουμε να συγχαρούμε την κυρία Χίρς. Ε, είναι πολύ καλή η δουλειά της. Ήταν πολύ επικοδομητική, πολύ δεκτική σε ό,τι αφορά τις δικές μας απόψεις. Η κυρία Ρενιέ μου λέει ότι 14, 133 και 124 ε, ε, έγιναν δεκτές. Ε, δύο μόνο θέματα μένουν εκρεμή Ενδεχομένως θα... Ε, θα μπορούσαν, να, να, θα μπορούσαν τελευταία στιγμή να ρυθμιστούν, αλλά στις ε, συμβαστικέ τροπολογίε Β και Μ και Σ, Β και Γ δεν μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Πάντως ε, είναι πολύ καλό, που η, ε, είναι πολύ καλό η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα των εργαζομένων και το νομικό πλαίσιο το οποίο απορρέει από, τις, από την νομοδότησή μας. Κυρία Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πραγματικά εξαιρετική εργασία της και τη συνεργασία που πέτυχε και πώς υιοθέτησε, πώς, πώς χειρίστηκε τις ε, πολλές επιφυλάξεις ε, ε των συναδέλφων ε, ε, και, και τελικά πέτυχε τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Από την πλευρά της δικής μου ομάδας πιστεύουμε ότι η ουσία του κανονισμού, ο στόχος ε, του κανονισμού είναι να προσφέρει περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την επεξεργασία και το χειρισμό όλου αυτού του θέματος των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο κανονισμός συμπεριλάβει βάση του άρθρου 82 ε, ένα κεφάλαιο για την απασχόληση θα πρέπει να μην είμαστε υπερβολικά ε, κανονιστικοί, να μην δηλαδή υιοθετήσουμε υπερβολικές κανονιστικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να ε, επιβαρύνουμε περισσότερο το άχθος της, ε, το κανονιστικό και τη γραφειοκρατία. Πιστεύω ότι πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν μια, ένα νομοθετικό πλαίσιο που λειτουργεί ικανοποιητικά ε, και πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός δεν επιδιώκει να περιορίσει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή του δικού τους κανονιστικού πλαισίου. Βεβαίως συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ψηλές ε, προδιαγραφές υψηλού επίπεδου και να ε, βοηθήσουμε βεβαίως να κατανοήσουν σαφέστρα τις διατάξεις αυτές άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη νομοθεσία. Υπάρχουν, υπάρχουν ένα-δύο συμβιβαστικοί τροπολογίε, τροπολογίες, ιδίως η τελευταία, το K, που δεν νομίζω να μπορούμε να υποστηρίξουμε. Είναι ε, πολύ περιοριστική, ιδίως η τελευταία παράγραφος D, δέλτα που αναφέρει το τηλέφωνο, τα email, το διαδίκτυο κλπ. για την αποφυγή απάτης. Όσον αφορά την συμβαστική F, δεν νομίζω. Δεν είναι θέμα αυτό της, απασχο... της Επιτροπής Απασχόλησης. Πρέπει αυτό να το χειριστεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Άλλες παρεμβάσεις. Αν όχι θα δώσω το λόγο στην κυρία, στην συγκεκριά μας. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε θα ψηφίσουμε αύριο πάλι και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τον Απρίλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, θέσεις μας. Τελειώσαμε το σημείο 11. Περνάμε στο 12. συμβαστικές τροπολογίες για την έκθεση Σόγκορ Ευρωπαϊκές Δημογραφικές Στατιστικές. Έχετε το λόγο. Thank you. I will speak in Hungarian. Θα μιλήσω στα ογκρικά, αν μου επιτρέπετε. Κυρίε και κύριοι, φαίνεται σαν είναι τεχνική αυτή η έκθεση, έχει ε, αυτή την μορφή, χρειαζόμαστε ε, σαφή και ακριβή κριτήρια ε, για τις δημογραφικές μας στατιστικές. πιστεύω ότι τα έγγραφα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις και σε μη τεχνικά θέματα. το Συμβούλιο ασχολείται με το ζήτημα αυτό από το 2010. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολιτικές, κοινωνικές και άλλου τύπου. Μπορεί να εξαρτάται ακόμα και το ευρωπαϊκό πνεύμα από αυτές. Η Ανατολική Ευρώπη, οι Βαλτικές χώρες, η Γερμανία, η Πορτογαλία ε, μπορεί να ε, δουν πολύ σαφώς αυτές οι επιπτώσεις. 57 τροπολογίες κατατέθηκαν, μία αποσύρθηκε. Ο στόχος είναι σαφής, χρειαζόμαστε δημογραφικούς, ενιαίους δημογραφικούς ε, δείκτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Πώ θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι δείκτες όμω αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, αυτή η απάντηση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ήδη ε, σε μία επιτροπή έχει γίνει ψηφοφορία και ε, στη δική τους νομοδότηση ε, αναφέρεται ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι για να υπολογιστεί ο αριθμός των διαμονών σε μια χώρα. Η Κομισιόν θα ε, διαθέτει στα χέρια της ε, θα διαθέτει στα χέρια της και άλλες μεθόδους λοιπόν. Ε, το Συμβούλιο βέβαια τελικά θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία και ελπίζω ότι θα επικρατήσει το συνολικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινό μας συμφέρον, με ελεγγύη από όλους προς όλους. Έχω κάποιες ανησυχίες για τους ορισμούς, για παράδειγμα στο τμήμα 2 και το τμήμα 3 ε, θα πρέπει να τους ξαναδούμε. Επίσης σε ό,τι αφορά το άρθρο 4 αν δούμε τα δύο πρώτα θέματα νομίζω χρειαζόμαστε ε, ε, διεθνή πρότυπα αν δείτε όμως το άρθρο 4 εκεί έχουμε σημαντικά προβλήματα πρέπει είναι σημαντικό να θυμηθούμε τη λογική που μόλις ανέφερα και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν έχουν μια μόνιμη κατοικία και αυτό το κείμενο θα τους επηρεάσει. Υπάρχουν σημαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις που θα πετύχουν ή θα αποτύχουν ε, σε συνάρτηση με το τελικό αποτέλεσμα της ε, πρότασης αυτής. Το κείμενο λοιπόν θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ε, θα επηρεάσει και τα μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένας ε, κανόνας προτιμησιακός. Επίσης, το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο λόγω της οικονομικής κρίσης γιατί έχουμε πολλές μετακινήσεις πληθυσμών τα στατιστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, χρειάζεται όμως να βασίζονται σε, ένα, σε μια ενιαία βάση. Και πρέπει να δούμε και το πώς θα χρησιμοποιηθούν. Ε, δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε ορισμένα πράγματα. Ορισμένες χώρες χάνουν πληθυσμό, ορισμένων αυξάνουν τον πληθυσμό λόγω της κρίσης και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, το ζήτημα είναι επίμαχο, λέει η Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν συμβαστικές τροπολογίες ακόμα. Θα δώσω το λόγο στην Αγγίνα Μπάστος και μετά στην κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή. Ε, με πολλή νυφαλιότητα αντιμετωπίζει το θέμα, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του. Το ζήτημα είναι σημαντικό και ευαίσθητο πολιτικά. Οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι πολύ σημαντικές σε ορισμένα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία είναι ένα από αυτά τα μέλη, ε, τα οποία μπορεί να πληγούν από την έκθεση αυτή αν δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για να αποφύγουμε τέτοιου είδους αρνητικές επιπτώσεις, ε, υπέβαλα κάποιες ε, προτάσεις τροπολογίας τις οποίες συνυπέγραψαν και άλλοι συναδελφοί του ΕΛΚ. Ε, για παράδειγμα ο κ. Ξάμπα. Ε, θα χρειαστεί ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο από το 2014 και μετά. Οι ψήφοι ε, αυτές θα πρέπει να καθορίζονται με βάση ε, τον αριθμό των ατόμων που έχουν μόνιμη κατοικία στο κάθε κράτος. Όχι συνήθις κατοικία, αλλά μόνιμη κατοικία. Και να μιλήσουμε για τον πληθυσμό των πολιτών, αριθμό των πολιτών. Αυτός ο ορισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι... Ε, ε, επηρεάζει τις χώρες ε, οι οποίες υφίστανται σε σημαντικές μεταναστευτικές ε, ροές για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους. δεν θα πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη αυτοί, αυτοί οι λόγοι γιατί οφείλονται στην οικονομική κρίση και δεν είναι δυνατόν να μειώσουν το βάρος της ψήφου κάθε χώρας ή τον αριθμό των ευρωβουλευτών που την αντιπροσωπεύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ο εισηγητής να τα καταφέρει, ε, διότι το δικό του κείμενο είναι πιο ισορροπημένο από την σημερινή φυστάμενη πρόταση. Ευχαριστώ. Από έκπληξη έκπληξη περνάω, λέει η κυρία Μπερές, γιατί από όταν ε, τέθησε εφαρμογή η συνθήκη της Αβώνας, ε, τροποποιήθηκε τουλάχιστον τρεις φορές και κανένα κράτος μέλος ποτέ δεν αμφισβήτησε τον κανόνα των ψηφοφοριών, τη στάθμης του ψήφου δηλαδή, της Λισαβόνας. Μέσω ενός κειμένου για στατιστικές να αμφισβητείται αυτό που τα κράτη-μέλη δέχτηκαν και στην είσοδό τους στην ένταξη της Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω της συνθήκης Λισαβόνας δεν μου φαίνεται μια καλή πρακτική. Η κυρία Παπαδοπούλου και μετά η κυρία Χάρκιν. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ σημαντικός φάκελος με πολλές αντιφατικές πτυχές και συζητήσαμε επί μακρόν το θέμα αυτό της ειδική πλειοψηφίας που ανέφερε η κυρία Μπάστος. Εγώ πρότεινα μία τροπολογία διότι πράγματι Υπάρχουν μεγάλες επιφυλάξεις από τον εισηγητή ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, κεντρικοευρωπαϊκές χώρες, επηρεάζονται κλπ. Αλλά είναι μια έκθεση τεχνικής ε, φύσης και είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες που θα παρασχεθούν από τα 27 κράτη-μέλη για να μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Διότι πολλές φορές είδαμε στο παρελθόν ότι δεν υπήρχε συνέπεια στις διαδικασίες, δηλαδή στη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών και εάν συγκρίνεται τις διαδικασίες από μία χώρα στην άλλη διαφέρουν σημαντικά. Είναι λοιπόν σημαντικό να επιτύχουμε συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες για αυτό το ντοσιέ. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο θέμα στο οποίο υπάρχουν αντιφατικές απόψεις. Ο εισηγητής δυστυχώς έκανε την προσπάθεια να εισαγάγει ένα ε, μεγάλο αριθμό ε, όρων, ορολογίες δηλαδή εκτεταμένες ορολογίες. Μιλάει για νέες περιφέρειες, new regions. Αυτό δεν συνάδει με τη διεθνή αποδεκτά ορολογία. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν ε, διεξάγει ε, ε, ενδελεχείς συζητήσεις με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να δεχθούμε καμία αλλαγή ορολογίας και ορισμών στο άρθρο 2 ούτε να επιτρέψουμε την εισαγωγή του όρου citizenship ηθαγένεια, αλλά να τηρήσουμε τη διεθνή ορολογία, τους διεθνούς ορισμούς. Τώρα ο στόχος αυτού του κανονισμού άρθρο 4 δεν θα πρέπει να ε, διαφοροποιήσουμε και εκεί τους όρους της ηθαγένειας ε, και δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του κυρίου Σόκορ αν δεχτούμε πολλές από τις προτάσεις του κυρίου Σόκορ θα υπάρχει αλυσιδωτή αντίδραση σε άλλους κανονισμούς διότι επαναλαμβάνω ότι προτείνει ορισμούς που δεν είναι αποδεκτοί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλούς άλλους κανονισμούς της Κομισιόν, από, από πλευράς Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν, ως σκιώδης εισηγήτρια, έχω υποβάλει τέσσερις συμβαστικές τροπολογίε τις οποίε έχουμε συζητήσει και με τους άλλους και του συζητητές και πιστεύω για να ολοκληρώσουμε αυτό το φάκελο σας παρακαλώ θερμά να μελετήσετε προσεκτικά τις τροπολογίες διότι ξέρω ότι μέσα στο ΑΕΚ υπάρχουν αντιφατικές, αντίθετες απόψεις δεν είναι ενωμένο στην ε, αξιολόγηση αυτών των τροπολογιών το ΕΛΚ. Δεν έχει μία μόφωνη άποψη. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ και από τον εισηγητή να ξανασκεφτεί αυτά τα οποία λέω. Ε, πρέπει να δεχτούμε την, τους ορισμούς του ΟΗΕ. Δεν μπορούμε εμείς ξαφνικά να παρουσιάσουμε νέα ορολογία, νέους ορισμούς. Και επίσης ε, να σας παραπέμπω στις βασικές τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Πιστεύω θα πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς από τους κέντρους ηγητές και για να επιτύχουμε μία, ε, ε, ένα συμβιβασμό. Η κυρία... Κυρία Μπάστος, μην προσπαθείτε να πείστε την κυρία Μωρέν Σαρτιέ με αυτόν τον τρόπο. Η κυρία Χάρκιν και μετά ο κύριος Σωρή. Ευχαριστώ. Λέει ναι, κυρία Χάρκιν, αντιφατικό έγγραφο αυτό, αντιφατικό ντοσιέ, ενώ ότι χρειάζονται συνεπείς και συνεκτικές στατιστικές. Ε, τα πράγματα δεν είναι διόλου απλά. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε όσο μπορούμε πιο πιστοί στο κείμενο του Συμβουλίου. Έχουμε λάβει ε, τις τροπολογίες από τους σοσιαλιστές και πιστεύω ότι γενικά μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Ήθελα να σχολιάσω το άρθρο 2 παράγραφος 1 υπο, ε, παράγραφος Δ υπό 2. Όσον αφορά τον ορισμό της συνήθους κατοικίας. Η πρόταση των σοσιαλιστών είναι ότι η συνήθις διαμονή είναι όπου είναι το μέρος όπου ο κάτοικο περνάει το περισσότερο χρόνο του, παρόλο που μπορεί σε ορισμένε περιόδους να λείπει, να είναι αλλού. Τώρα, ε, τα δημογραφικά στοιχεία του 2008-2009 ε, ορίζουν τι σημαίνει προσωρινή απουσία. Προσωρινή απουσία, διαλόγους, α, β, γ κλπ παραδείγματο χάρη προσκυνήματος. Όταν διάβασα όλα αυτά τα παραδείγματα, έκρινα ότι ήδη αυτά καλύπτονται από τον κανονισμό του 2008. Γι' αυτό λοιπόν, για λόγους συνέπειας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στην κοινή ορολογία δεν ε, είναι τίποτα το ριζοσπαστικό το οποίο ε, προτείνω και νομίζω ότι έτσι μπορεί να περάσει η τροπολογία. Το άλλο που μας αφορά ιδιαίτερα είναι η χρονική διάρκεια στην οποία διαμένει στη συνήθεια κατοικία του ένα άτομα και ο, κύριος, ο εισηγητής προτείνει πέντε χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο που προτείνουν 12 μήνες είναι καλύτερη πρόταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση του εισηγητή. Ξέρω, ο κ. Σόγκορ το πρότεινε τα 5 χρόνια, αλλά από ό,τι ξέρω εγώ και παρακαλώ διορθώστε με, αυτή η πενταετής περίοδος δεν εμφανίζεται πουθενά, πουθενά σε κανέναν άλλον διεθνή ορισμό που χρησιμοποιείται και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να ε, παραμείνει ενισχύ ε, η περίοδος των 12 μηνών όπως πρότεινε η Κομισιό και συμφώνησε το Συμβούλιο. Επίσης, και πάλι εδώ αναφέρουμε στις προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες των σοσιαλιστών μπορούμε να συμφωνούσουμε με τη συμβαστική 4 που αφορά την μη διάκριση αναφύλω. Ο κύριος Σωρή. Θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω στα όσα είπατε εσείς, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι κανείς ε, αμφισβητεί τους μηχανισμούς λήψη απόφασης ε, που υιοθετήθηκαν μέσω της Σύνθηκης της Λισαβόνας. Μιλάμε για έναν στατιστικό μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να ε, γνωρίζουμε πόσα άτομα βρίσκονται κάθε στιγμή στην επικράτεια κάποιου κάθε κράτους μέλους. Για δημογραφία μιλάμε, όχι για τίποτα άλλο. Η δημογραφία βέβαια καθορίζει την ε, στάθμιση των ψήφων. Τώρα, ε, εγώ σέβομαι πολύ τους στατιστικολόγους, έχω συνεργαστεί μαζί τους για αρκετά χρόνια και γνωρίζω λίγο πολύ πώς λειτουργούν τα στατιστικά, έχω εμπειρία. Τώρα, ας δούμε λίγο τους ορισμούς η συνήθις διαμονή, πώς καθορίζεται, πώς χρησιμοποιείται αυτή η έννοια κλπ. Να σας πω δύο λόγια για αυτό το ζήτημα, αν μου επιτρέπετε. Οι 12 μήνες είναι πολύ μικρή περίοδος κατά την άποψή μου. Δεν μιλούμε για μια καινούργια διαδικασία. Οι στατιστικές χρησιμοποιούν αυτό τον όρο εδώ και πολύ καιρό. Η συνήθις διαμονή είναι ο όρος που χρησιμοποιείται και η περίοδος αναφοράς ε, στο παρελθόν ήταν 10 χρόνια. Συνήθως ε, οι απογραφές γίνονται κάθε 10 χρόνια και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται αυτή η περίοδος ως βάση. Μην ξεχνάμε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη οι στατιστικά συλλέγονται κάθε χρόνο. Οπότε η Κομισιόν, αν καταλαβαίνω καλά το στόχο της, είναι να ε, εξυγχρονίσουν τα κείμενα έτσι ώστε όταν έχουμε ετήσια στατιστικά στοιχεία σε ορισμένε χώρε, αυτά τα στοιχεία να εντάσσονται στο συνολικό υπολογισμό αμέσω. Η Κομισιόν θέλει να επιταχύνει λοιπόν τα πράγματα. Να μην καθυστερούμε δύο χρόνια, αλλά ένα χρόνο. Καταλαβαίνω αυτό το στόχο, καταλαβαίνω αυτή την πρόθεση. Αυτό που δυσκολεύομαι να κατανοήσω όμω είναι το εξή. Η διαμονή, ε, μάλλον ο συνήθω διαμένων ε, χρειάζεται να υπάρχει κάποια δέσμευση μεταξύ αυτού του ατόμου και της χώρας στην οποία συνήθως διαμένει. Πολλές φορές μπορεί να μιλάμε για άτομα που διαμένουν μακριά από τις οικογένειές τους και να έχουν ε, υποχρεώσει κάπου αλλού. Μπορεί αυτά τα άτομα να γυρίζουν σπίτι τους συχνά. Ε, το κάνω εγώ, για παράδειγμα, ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουγγαρία. Το γνωρίζω πολύ καλά. Και ξέρω και πολλούς άλλους, Ισπανούς, Ιταλούς και άλλους ανθρώπους που είναι, ε, που κινούνται πάρα πολύ συχνά μεταξύ δύο χωρών. Συνεπώς, δύο, 12 μήνες είναι μικρότεροι από μια συνήθι εργασιακή σύμβαση. Ε, μια εργασιακή σύμβαση συνήθως διαρκεί 3-4 χρόνια. Το γεγονός ότι έχεις μια τέτοια σύμβαση δεν σε κάνει Βέλγο παρόλο που είσαι Ρουμάνος, Ούγκρος ή οτιδήποτε άλλο εργάζεσαι ενδεχομένω στι Βρυξέλλε, έχει μια εργασιακή σύμβαση στι Βρυξέλλε. Αυτό δεν σε κάνει Βέλγο. Μετά, επιχειρήσει στέλνουν του εργαζόμενου του σε άλλη χώρα ε, για κάποια χρονικά διαστήματα. Συνεπώ, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ε, δεν συμφωνώ με την Μάριον ότι ε, η έννοια των πέντε ετών δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Η μόνιμη κατοικία, η μόνιμη κατοικία από την άλλη μεριά, σχετίζεται με άλλη σύμβαση, η οποία μιλά για πέντε χρόνια ή μιλά για μια διάρκεια πέντε ετών. Αλλά δεν μιλούμε για μόνιμη κατοικία αυτή τη στιγμή. Μιλούμε για άτομα τα οποία σύμφωνα με την πρόταση διαμένουν σε άλλη χώρα τουλάχιστον ένα έτος. Τουλάχιστον ένα έτος. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή περίοδος αναφοράς, όχι τα πέντε έτη. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Συζητήσαμε τα στατιστικά, τη φύση των στατιστικών, κλείνω αυτή την παρένθεση. Στο Συμβούλιο δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα για αυτό το ζήτημα. Οι χώρες έστειλαν εμπειρογνώμονες, στατιστικολόγους, εξέτασαν την πρόταση και έκανε και κάποιες προτάσεις. Όλοι συμφώνησαν επί τεχνικού επίπεδου και γι' αυτό το λόγο και οι κυβερνήσεις συμφώνησαν. Εν τω μεταξύ βέβαια υπογράφηκε η συνδίκη της Λισαβόνας, Ξέρετε ότι η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ παλιά και η συνθήκη της Αβώνας έχει συγκεκριμένε επιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε σχέση με τη στατιστική μέθοδο, μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιούμε. Και το Κοινοβούλιο άρχισε να υψώνει τη φωνή του γιατί αρχίσαμε να αμφισβητούμε τη μέθοδο. Είπαμε ότι υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν είχαμε προβλέψει δεν αμφισβητούμε την εμπειρογνωμοσύνη των στατιστικών λόγων μας. Απλά λέμε ότι όταν έκαναν τους υπολογισμούς τους, ίσως δεν έλαβαν υπόψη αυτά τα οποία λαμβάνουμε εμείς υπόψη, δηλαδή το, το, τη χρήση, την ε, εκ των υστέρων χρήση αυτών των στατιστικών στοιχείων. Για παράδειγμα, επιπτώσεις σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης, αποφάσεων. Δεν ξέρω αν σκέφτηκαν το Συμβούλιο, την Κομισιόν, δεν είδα ποτέ ένα μοντέλο που να υπολογίζει ε, τις επιπτώσεις αυτού του κειμένου στο μηχανισμό λήψη αποφάσεων, πώς ε, θα μπορούσε να διαστρεβλωθεί να αλλοιωθεί ε, η στάθμιση της ψήφου κλπ. Είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Δεν είναι σαφές. Είναι κάτι που θα έπρεπε να λάβουμε σοβαρά υπόψη, είναι σημαντικές επιπτώσεις, θα έπρεπε να υπολογιστούν. Θα έπρεπε δηλαδή να δούμε, ε, έχουμε 100.000 άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτή τη χώρα αλλά καταμετρώνται κάπου αλλού. Αυτό θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην στάθμιση ψήφου. Δεν ξέρουμε, πρέπει να, πρέπει να υπολογιστεί. Αλλά μπορεί και ένα μικρότερο νούμερο να είχε επιπτώσεις. Δεν έχουμε δει παραδείγματα. Αν βλέπαμε παραδείγματα τότε πράγματι θα είχαμε κάτι να σκεφτούμε, να βασιστούμε πάνω του. Ε, προτάθηκαν τα πέντε έτη. Δεν ξέρω Ίσως είναι καλή ιδέα. στον τριμερή διάλογο θα το συζητήσουμε, θα ανταλλάξουμε επιχειρήματα και ίσως θα ακουστούν και πιο πιστικά παραδείγματα ε, απτά. Έτσι ώστε να πιστούμε ότι αυτή η α ή β μέθοδος δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το α, β ή γ κράτος μέλος. Θα υποχρεώσουμε το Συμβούλιο να μας αποδείξει ε, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα στην πράξη, ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης στην πράξη. Και έτσι θα βάλουμε και τελεία και παύλα στη συζήτηση. Αυτά είναι τα δικά μου σχόλια. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να σκεφτεί, να προβληματιστεί για τον πολιτικό του ρόλο. Ευχαριστώ αρχίζει να μας περιορίζει ο χρόνος. Δεν μπορώ να ακούω ομιλητέ οι οποίοι μιλούν τρει φορέ περισσότερο από τον εισηγητή. Σα παρακαλώ καθένα να αυτοπεριορίζετε και να αυτοπιθαρχείτε. Η Ούμαν Ρόιτερ. Όχι, όχι, πρώτα ένα άλλο ομιλητή. Πώ θα. Ο κύριο Ούγκου Ρεάνου. Λοιπόν, ότι έχουμε, έχουμε διαφορετικά στατιστικά στοιχεία. Ε, υπάρχουν οι έννοιες όπως η συνήθις διαμονή. Αυτό είναι συνταγή για αναξιόπιστα, χαοτικά, στατιστικά στοιχεία. Αν κοιτάξετε το άρθρο 2 που μιλάει για τη συνήθεια κατοικία και την 12 περίοδο. Η βάση αυτής της έννοιας είναι ότι κάποιος προσμετράται αν βρεθεί κάπου για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι. Περί αυτού πρόκειται. Είναι όμως μια αόριστη έννοια. Εφιστώ την προσοχή των συναδέλφων, λοιπόν, στις τροπολογίες 8 και 9 του εισηγητή και ζητώ να τις υποστηρίξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Όιμαν Κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη πρόταση που ακούστηκε κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση του ΑΕΛΚ με αποσταθεροποίησε λιγάκι, γιατί εμπεριέχει κάποια σημεία που κατά την άποψή μου δεν έχουν θέση σε μια αξιοπρεπή Ευρώπη. Υπάρχει μία τροπολογία για την εθνότητα. Ευτυχώς δεν τη δέχεστε. Χάρηκα γι' αυτό. Και υπάρχουν διάφορες έννοιες οι οποίες είναι λίγο προβληματικές. Η ηθαγένεια, το citizenship. Σε αυτή την περίπτωση θα σήμαινε ότι οι Ιρλανδοί και οι Ιταλοί είναι τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη, γιατί ο πληθυσμό τους είναι ο πιο εξαπλωμένος στην Ιφίλιο. Δεν νομίζω ότι έχει έννοια αυτή, έχει νόημα αυτή η έννοια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε χωρίς να βασιστούμε στατιστικές είναι να ε, προκύψουν και κάποιες πολιτικές συνέπειες, τις οποίες θέλουμε να εξετάσουμε. αν λάβουμε υπόψη μα την ειδική πλειοψηφία για τι ε, συνέπειε αυτέ, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί αν, αν παρασπούμε του κατοίκου των κάτω χωρών, 6,5 εκατομμύρια, 12 μονάδε για αυτού. Μετά, Ρουμανία, 21 εκατομμύρια. 13 σημεία. Ακόμα και αν θα ήθελα να το επηρεάσω αυτό με μια πολιτική διάσταση, με αυτά τα νούμερα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν βάλουμε, λάβουμε υπόψη μας αυτή την πενταετή περίοδο, τι κάνουμε με αυτά τα άτομα τα οποία μένουν πέντε χρόνια στην άλλο κρατός μέλος. Γιατί επί πέντε χρόνια αυτά τα άτομα καλύπτονται από το κράτο, κράτος μέλος διαμονής τους. Αυτό τα αναλαμβάνει, αυτό είναι υπεύθυνο για αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν τις, τις δημόσιες μεταφορές, τα νοσοκομεία, ε, τη στέγαση. Όλα αυτά επιδοτούνται. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα πέντε χρόνια δεν λαμβάνουν υπόψη. Και θα εξετάσω επίσης και τους συμβασμούς όπως έχουν προταθεί και θα εξετάσω και το, και το κείμενο του Συμβουλίου, το οποίο έχω ήδη δει μία φορά. Και με βάση αυτά όλα τα στοιχεία θα επιλέξω τη στάση μου. Αλλά το πολιτικό επιχείρημα ότι... Και δεν ξέρω αν αυτό θα ε, Το πολιτικό επιχείρημα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πείσει τους συναδέλφους, αλλά αυτή είναι η απόψή μου. Εγώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις για αυτό το θέμα. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι δημογραφικές στατιστικές, όπως είπε και ο κύριος Σόρη, έχει αλλάξει. Το 19ο αιώνα κάναμε μία απογραφή κάθε 10 χρόνια και στέλναμε τους χωροφύλακες πάνω στα άλογα στα χωριά για να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στα σπίτια. Έκτοτε όμως άλλαξαν τα πράγματα. <clears throat> Και οι στατιστικές μέθοδοι ε, ευτυχώς μας επέτρεψαν να έχουμε καλύτερα στατιστικά στοιχεία. Όχι πάντα αρκετά, όχι πάντα πολύ ποιοτικά, γιατί θέλουμε να υπολογίσουμε πούμε, το κατόφλι φτώχεια και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να περιμένουμε καιρό για να έχουμε τους σωστούς, τα σωστά αριθμητικά στοιχεία. Αλλά στον τομέα της δημογραφίας, εκεί όλοι ξέρουμε ότι έχουμε σημειώσει πολύ πρόοδο. Τώρα, η έννοια αυτής της πρόοδου είναι να μπορούμε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα και στα εργαλεία, μάλλον τα εργαλεία στην πραγματικότητα. Απέναντι στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που αφορούν τη σύνθεση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο που οι στατιστικολόγοι επέλεξαν και επικύρωσαν την πρόταση της Κομισιόν. Γιατί είναι προτάσεις που είναι σωστές, βασισμένες σε στοιχεία, σε πραγματογνωμοσύνη. Ε, αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Το δεύτερο επιχείρημα, ο δεύτερος άξονας επιχειρημάτων είναι η διασύνδεση που κάνουμε ανάμεσα στον ορισμό τη ε, συνήθου κατοικία που υπάρχει στο άρθρο 2 και το πώ συνδέεται αυτό ε, ή μάλλον πώ αντιμετωπίζεται το ίδιο θέμα στο άρθρο 4. Νομίζω ότι στο άρθρο 4 υπάρχει ένα ορισμό που είναι πολύ πιο έτσι, εκλεπτισμένος θα έλεγα, γιατί αυτό το άρθρο συνδέεται με το θέμα της χρήσης των στατιστικών δεδομένων για να καθορίσουμε το ειδικό βάρος του καθενός, ε, με σκοπό την, της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. Ε, οι συμβαστικές προτάσεις των σοσιαλιστών ε, λαμβάνουν υπόψη τη διαιτερότητα των στατιστικών στο άρθρο 4 αν γίνει αυτό, που αν γίνει αυτό γενικός κανόνας για τον καθορισμό ε, των διαμενών των πληθυσμών, νομίζω ότι θα μας επέτρεπε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα πολύ καλό. Από την πρόταση της κυρίας Χάρκιν κατάλαβα ότι η κυρία Χάρκιν είναι ανοιχτή σε αυτή τη δυνατότητα. Μήπως... Ε, Υπάρχει ένα κείμενο του Συμβουλίου προϋπάρχων για τον ε, ορισμό της συνήθους κατοικίας που συμπεριλαμβάνει κατηγορίες που για μένα είναι εντυπωσιακέ. Ε, με καταπλήσουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται. Δηλαδή κάποιος ας πούμε πάει να κάνει ένα προσκύνημα ή να, κάνει, να λάβει μια θεραπεία ας πούμε σε ένα νοσοκομείο σε μια άλλη χώρα, λαμβάνεται υπόψη αυτό και αυτό μου φαίνεται ε, λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, αν χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μα όλα αυτά για να φτάσουμε σε συμβιβασμό, α, τι να πω, πρέπει να ακούσω και την άποψη των μελών τη Επιτροπής. Ο κύριος Τόμα Μαν που είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνήθως εμεί κάνουμε την προσπάθεια να συμφωνήσουμε. Παρακολουθώντας τώρα αυτή τη συζήτηση βλέπω την απόσταση, μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Δεν έχουμε ακόμα τις συμβιβαστικέ τροπολογίες και αν βλέπω πόσο διαφορετικές είναι οι θέσεις, ανησυχώ. Πιστεύω ότι η ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων μέχρι τις πρακτικές εφαρμογές, δηλαδή να κρίνουμε τώρα πότε είναι κάποιος ε, ηθαγενής, ε, ε, πότε είναι και πού η διαμονή, πόσα είναι η χρονική διάρκεια. Αυτά είναι όλα θέματα ερμηνείας. Θέλουμε τώρα να ψηφίσουμε όταν βλέπουμε τόσες αντίθετες και διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου έχουμε μία βάση ομόφωνη Έχουμε, έχουμε πολλές εκθέσεις όπου η βάση μας ήταν ε, ομόφωνη, ήταν ενιαία και εν συνεχεία διαμορφώσαμε διαφορετικά μερικές πτυχές. Αλλά εδώ εκπέμπουνε μηνύματα κινδύνου και γι' αυτό ρωτώ μήπως μπορούμε να αναβάλουμε, να απεξεργαστούμε την κοινή γραμμή, την κοινή θέση μας ε, δεδομένου, παρά να έχουμε διαφορετικές θέσεις και απόψεις από τις διάφορες ομάδες. Εσείς μιλήσατε ήδη πιο πολύ από κάθε άλλο σε αυτήν την συνεδρίαση. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε κείμενο από την ένα κείμενο από την ε, Κομισιόν που μας ε, διαβεβαιώνει όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία το εξής. Οι χώρες ενθαρρύνουν να υποβάλουν τα στατιστικά στις στοιχεία. Αν δεν είναι δυνατό να το κάνουν αυτό, υποβάλλουν τα στοιχεία του νόμιμου πληθυσμού. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς ε, πώς δίνεται αυτή η δυνατότητα διαφορετικών υπολογισμών. Στη μία περίπτωση δεν υπολογίζουν βάση της μεθόδου α και στην άλλη βάση της μεθόδου β. Ο Τόμας ε, ε, έθεσε το θέμα, διακόπτει η πρόεδρος Κοιτάξτε, θέλει, ο εισηγητής πρέπει να δώσει το λόγο να απαντήσει στι ανησυχίε σα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω την κυρία Παπαδοπούλου, θα τη δώσω το λόγο για μία στιγμή. Όχι κύριε Ορή, ε, ένα λεπτό κυρία Παπαδοπούλου ή δευτερόλεπτο. Θα είμαι πολύ σύντομη. Στην σύντομη εισαγωγή μου είχα πει ότι είχαμε έντονες συζητήσει με το Συμβούλιο και προσπαθήσαμε, κύριε Μαν, να φτάσουμε σε συμβιβασμό. Γιατί αν πάμε σε ψηφοφορία αύριο, πρέπει να δούμε ποιες πολιτικές ομάδες συμφωνούν και ποιες διαφωνούν. Τίποτα άλλο. Σας σταματώ. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, για να απαντήσω στον κύριο Όρη. Αυτή η απάντηση της Κομισιόν είναι ο συμβασμός υπαριθμών 3. Το δεχτήκαμε. Σας προτείνω, προτείνω στις πολιτικές ομάδες να διαβάσουν προσεκτικά. Θα το κάνουν, διακόπτει συνέχεια η Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, ζητά συγγνώμη ο υπεύθυνο διευθυντή για το θέμα, ο οποίο αναγκάστηκε να παραμείνει στο Λουξεμβούργο για ένα σοβαρό οικογενειακό του πρόβλημα. Α, ε, και επίση υπάρχει και ένα άλλο υπεύθυνο που είναι μπλοκαρισμένο ε, στο Ναμύρ αυτή τη στιγμή, γιατί υπήρχε, υπήρχε στάση τεχνικού πρόβλημα, δηλαδή με τον τρένο τεχνικού χαρακτήρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θεωρούμε ότι οι ανάγκες ε, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, είναι μια αρχή που τη δεχόμαστε. Και η αρχή που βασίζεται στην, ε, στον εθελοντισμό δεν ισχύει από την επόμενη περίοδο ψηφοφορία από το 2014. Όταν σκέφτηκε η Κομισιόν τι στάση θα πρέπει να έχει, ε, δεν προσπάθησε να ερμηνεύσει τις ε, συνθήκες. Τεχνικά προσπαθήσαμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να έχουμε ενιαίες ε, διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε όλα τα νούμερα μεταξύ όλων των κρατών μελών. Προσπαθήσαμε δηλαδή να σεβαστούμε τους άλλους κανονισμούς και κοινοτικά κείμενα που αναφέρονται σε δεδομένα πληθυσμών. Επίσης, Θέλαμε να λάβουμε υπόψη μα του ε, διεθνά συμπεφωνημένου ορισμού, ούτω ώστε να εγγυηθούμε μία αντικειμενικότητα στι αποφάσει. Τρίτον, προσπαθήσαμε να έχουμε κριτήρια τα οποία είναι σταθερά και μόνιμα συν το χρόνο, ανεξάρτητα από βραχυπρόθεσμε καταστάσεις. Οι στατιστικολόγοι ξέρουν ότι ο ορισμός των πληθυσμών, όπω είπε και η κυρία Πρόεδρο, ε, πάντα περιέχει περίπλοκα θέματα. Γι' αυτό η πρόταση που έχετε μπροστά σας είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς σειράς διαβουλεύσεων μεταξύ των ε, πυρογνωμών για τα στατιστικά που θεωρούν ότι η συνήθις κατοικία θα πρέπει να βασιστεί σε δεδομένα 12 μήνες διάρκειας και είναι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε ποιος είναι ο συνολικός πληθυσμός. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο καονισμός έχει δύο στόχους. Από την μία, να έχουμε ε, το συνολικό πληθυσμό με κάποια βάση και από την, να, άλλη να έχουμε δημογραφικά στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσουμε για εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Σε ό,τι αφορά τα νούμερα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το σύστημα ψηφοφορίας με δική πλειοψηφία, η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ορισμού συγκρίσιμου όλα τα κράτη-μέλη. Ακριβώς αυτό έχετε στο άρθρο που ζητάει από τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τη συνήθη κατοικία. Αυτό τον ορισμό όπως ε, ορίζεται με βάση τα άνωθη κριτήρια. Τώρα, για το θέμα του άρθρου 3, το θέμα που έθεσε ο κύριος Σόρη. Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία? Ναι, υπάρχει. Όντω, για τα νούμερα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις μεταβλητές που αφορούν τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής τα νούμερα που θα πρέπει να στέλνουν κάθε Σεπτέμβριο τα κράτη-μέλη για να δούμε ε, το νούμερο του συνολικού πληθυσμού είναι στοιχεία που έχουμε, έχουμε καλύτερη ευελιξία. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την πρότασή μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι κάναμε μια μακρά τεχνική προσπάθεια, ούτω ώστε να είναι όσο να τον πιο αξιόπιστα αυτά τα ε, νούμερα μεταξύ όλων των κρατών μελών και θεωρούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις μας στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου και εκεί είτε μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο είτε να σας δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος. Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη ψηφοφορία αυτή για αυτό το κείμενο. Το θέμα είναι αν οι πολιτικές ομάδες θέλουν περισσότερο χρόνο για να ετοιμάσουν συμβιβασμούς και να κοιτάξουν τις, συμβαστικέ, τις συμβαστικές τροπολογίες των σοσιαλιστών. Έχει νόημα αν υπάρχει έτσι ένα άνοιγμα πνεύματος. Αλλά φοβάμαι για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί, ειλικρινά σας το λέω, η παρουσίαση της Κομισιόν το αποδεικνύει ότι αυτές οι στατιστικές πρέπει να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε την 1η Ιανουαρίου του 2014. Δεν αποκλείεται το 1η Πρώτου του 2014 να υπάρχει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί και δεν μπορώ να προδικάσω, εν πάση όλα αυτά τα πράγματα. Όμω η διαπραγμάτευση μετά με το Συμβούλιο θα απαιτήσει και αυτή κάποιο χρόνο. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει εν συνεχεία να εφαρμόσουν το κείμενο. Οπότε, τι να κάνουμε. Θα προτιμούσα οι ομάδε να συμφωνήσουν το ταχύτερο δυνατόν. Ακόμα και αν χρειαστεί στη συνέχεια να πάμε στην Ολομέλεια προκειμένου να καθορίσουμε την εντολή διαπραγμάτευση. σω αυτή είναι η λύση διαφυγή. Κύριε Ωρή, θα σας ξαναδώσω το λόγο για λιγότερο από ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συμφωνώ σε αυτό υπό μία προϋπόθεση ιδέα αναβολής, με την ιδέα δηλαδή ότι θα γίνει μία αναβολή ε, ή θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε έναν ε, πρότυπο υπολογισμό, ένα μοντέλο υπολογισμού για να δούμε πώς, ε, τι επιπτώσεις θα έχει αυτός ο ορισμός και τι επιπτώσεις θα έχει αν γίνει δική ψηφοφορία με δική ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Πέστε μας λοιπόν τι θα γίνει. Μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ένας πολύ καλός υπολογισμός ή μπορεί να αποδειχθεί κακός. Η Κομισιόν έχει μια μελέτη επιπτώσεων, ε, ξέρει τα διάφορα σενάρια και έχει κάνει σχετική μελέτη επιπτώσεων. Όχι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να καθυστερήσουμε έξι μήνε τουλάχιστον, μην πω και ένα χρόνο. Ο κύριο Στέρκα. Καταλαβαίνω πολύ καλά το αίτημα του κύριου Τόμας Μαν. Όμως, η εμπειρία μας, μας λέει, μας διδάσκει ότι είναι μια συζήτηση που, τεχνική συζήτηση, στατιστική συζήτηση που κάνουν οι πολιτικοί. Αυτό θα μπορούσε να διονυστεί. Διότι ε, ίσως χρειαστεί να, πάμε, να γυρίσουμε στο, στα έδρανα του Πανεπιστημίου για να μάθουμε στατιστική εμείς πολιτική. Θα πρέπει... Δεν είναι δυνατόν οι υπάλληλοι να κάνουν δουλειά των πολιτικών και η πολιτική δουλειά των υπαλλήλων. Πολύ δε περισσότερο σε ένα κλάδο όπως η στατιστική που έχει τις ιδιαιτερότητές της. Έχει μια ιστορία αιώνων. Πώς είναι να το να συζητούμε για θέματα στατιστικά μεταξύ μας. Εγώ εμπιστεύομαι τους ειδικούς. Συνεπώς τα τεχνικά θέματα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητό μας. Και το θέμα αυτό είναι πραγματικά πολύ τεχνικό. Το έχουμε συζητήσει σε όλες του τις πολιτικές διαστάσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε γιατί έτσι λύνονται πολιτικά τα ζητήματα. Αλλιώς πιστεύω ότι θα ε, καθυστερήσουμε παόριστον. Πρόεδρος, διατηρούμε το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη και θα δούμε πώς θα οριστεί η ε, εντολή, η εντολή Ε, θα έρθει στη μέση διάταξη αύριο το θέμα. Τελειώσαμε με το 12. κύριε Σιγητά, θέλετε το λόγο. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Χάρκιν και στην κυρία Παπαδοπούλου εν συντομία. Είπα προηγουμένως ότι ε, το θέμα δεν αφορά μόνο την Ανατολική Ευρώπη. Όχι, δεν αφορά μόνο την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, ε, να σας πω ότι μπορούμε να δεχτούμε τους, ε, τις προτάσεις για τους ορισμούς της σοσιαλιστικής ομάδας. Έχει κάποιες τροπολογίες η σοσιαλιστική ομάδα. Μετά, ε, προς την κυρία Χάρκιν, να πω το εξής. νομίζω ότι οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν τα πέντε χρόνια αναφέρονται στην οδηγία σας, που, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Σωρή. Πρόεδρος, ακούσαμε τις ε, παρατηρήσεις του εισηγητή, θα ψηφίσουμε αύριο. Πριν περάσουμε στο σημείο 13, θα ήθελα να επανέλθω στο 2, να καλωσορίσω τον, τον Τζόναθαν Μπουσούτιλ και τον Νίκολα Τρόσ και οι δύο εθνικοί ε, εμπειρογνώμονες, όχι, βοηθή της ε, Γραμματείας της Επιτροπής από 1η Φεβρουαρίου. Α σηκωθούν, ε, παρόλο που ξέρω ότι είναι λίγο ντροπαλοί, α σηκωθούν να τους χαιρετήσουμε. Ωραία, καλώς ήρθατε. Βοηθή, καινούργη βοηθή στη γραμματεία μας. Dank, äh, Ο κύριος Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ε, ενημερώσω για τις υπηρεσίες εδάφους. Είχαμε μία με συνάντηση την, τελευταία, την περασμένη Δευτέρα και δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για μία περαιτέρω συμβιβαστική λύση. Θέλω να πω ότι οι τέσσερις τομείς, οι τέσσερις κατηγορίες που έχουμε, όπου που περιορίζεται η πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να διευρυνθούν σε 11. Ε, συζητήσαμε πολλές συμβαστικές προτάσεις και στις Βρυξέλλες και στην επίσκεψή μας ε, στο, στη Φραγκφούρτη και στο Βερολίνο, ιδιαίτερα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και λόγω της ημέρας αυτής προσπαθήσαμε πράγματι να συνεργαστούμε αρμονικά. Ε, διαπιστώσαμε όμως δυστυχώς ότι δεν το καταφέραμε αυτό, να συμφωνήσουμε δηλαδή απολύτως και να καταλήξουμε σε συμβιβαστική λύση. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε, διοργανώσουμε μια δεύτερη συνάντηση πριν από τη συνεδρίασή μας με τους Κιώδης, αλλά ε, θέλουμε να επιτύχουμε αυτά τα οποία αποφασίσαμε μαζί στον τελευταίο συμβιβασμό να το, διατηρήσουμε για την Επιτροπή Μεταφορών. Η Επιτροπή Μεταφορών περιμένει την ψηφοφορία της Επιτροπής Απασχόλησης και θέλουμε αύριο να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας. Όχι σε κάθε πτυχή και λεπτομέρεια της έκθεσης. Θέλουμε όμως να διατηρηθεί αυτή η έκθεση ζωντανή για να δώσει ένα μήνυμα στην Επιτροπή Μεταφορών διότι στην Ολομέλεια θα πρέπει να αποφασίσουμε τελικά. αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να υπονομευθεί η δική μας στάση, διότι το, η πρόταση αυτή αφορά πάρα πολλά κοινωνικά μέτρα για τους απασχολούμενους. Αυτός ο κίνδυνος υπονόμευσης είναι πολύ μεγάλος και γι' αυτό θέλουμε να φροντίσουμε ε, να συζητηθεί οπωσδήποτε αύριο και να ψηφιστεί και να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι ο συμβιβασμό μας διατηρείται, είναι ζωντανός και ισχύει και δεν φεύγει από την ατζέντα. Επίσης ήθελα να προτείνω μήπως ε, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε λίγο χρόνο έτσι ώστε ε, δεδομένου ότι δεν βλέπω πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις απόψεις μας αυτό το μήνα ακόμα και στην επιτοπή Μεταφορών οι απόψεις είναι διαφορετικές ε, και αντιφατικές. Ε, γι' αυτό θα έλεγα να κερδίσουμε ένα μήνα ακόμα. Θα ήθελα όμως αύριο να επιβεβαιώσετε ότι ο δικός μας, η δική μας συμβαστική πρόταση ισχύει και αυτό θα πρέπει να το δηλώσουμε σαφέστατα στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά αυτούς που εργάστηκαν έντονα και Ίσως θα μπορούσαμε τελικά να καταλήξουμε ε, σε μια συμβιβαστική λύση, αλλά δεν μπορέσαμε να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω σε αυτά τα οποία είχαμε επιτύχει μαζί. Ε, καλή βούληση δεν έλειπε, υπήρχε πάντοτε, αλλά δεν καταλήξαμε να, σε, σε κάποιο άλλο θετικό πρόσθετο στοιχείο. Η κυρία Χίρς. Δίνω τώρα τον λόγο στην Γιούτα Στάνμπρουκ, στην ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να διαπιστώσω ότι οι επιπτώσει στο άνοιγμα της αγοράς στους εργαζόμενους δεν είναι καθαρά γερμανικό πρόβλημα. Οι επιπτώσεις αυτές συζητήθηκαν και ε, λεπτομερώς ε, και συχνά τον περασμένο χρόνο. Είναι γεγονός ε, όταν δίνονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων περιφερειών στον κόσμο και όταν τέτοια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δεν μπορούν να τα κερδίσουν οι δικές μας εταιρείες εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστική μας θέση με ποιότητα και ασφάλεια. Αυτό το πακέτο, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του συζητείται στην Επιτροπή Μεταφορών, δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις ε, αυτή τη στιγμή εκφράζω μια μεγάλη ανησυχία, ακόμα και μεταξύ των συναδέλφων της Επιτροπής Μεταφορών, το τι γίνεται δηλαδή στους ουρανούς. Εμείς θέλουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία προ όφελο των εργαζομένων, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις χειρότερες εξελίξεις, τις χειρότερες επιπτώσεις. Οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί αντιτίθενται σε κάθε πρόταση ε, ε, απελευθέρωσης. Ελπίζω αυτό να μην περάσει, αυτή η πλήρης αντίθεση σε όλα τα οποία είναι κατά της απελευθέρωσης. Ε, επίσης οι φιλελεύθεροι και αυτοί ανησυχούν και αυτοί επιθυμώ να αποδυναμώσουν ε, τα μειονεκτήματα για τους εργαζόμενους. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν θέλουμε να φυγούν ε, ε, οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους και να πέσουν σε δυσμενέστερη θέση. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό. Αλλά στην τελευταία ψηφοφορία, ενώ η καρδιά μου έλεγε να καταψηφίσω, ε, δεν το έκανα για να αποφύγω τυχόν ε, χειροτέρευση της κατάστασης των εργαζομένων. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα συμβασμό εάν σε κάποια ε, εξαγορά ενημερωθούν και συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Έχω και νομικά προβλήματα σε αυτό το σημείο. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν εργαζόμενοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην ίδια επιχείρηση. Εμείς ως σοσιαλιστές και δημοκράτες θα, μπορέσουμε θα, θα αναγκαστούμε δυστυχώς να συμφωνήσουμε στο λιγότερο κακό, στο, στο μη δηλαδή. Ε, ε, ο κύριος ε, Μπαχ. Ε, είμαι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών ε, και γι' αυτό ήθελα να μιλήσω, δεδομένου ότι συνεργάστηκα και ασχολήθηκα και είμαι ενημερωμένος ε, για τις διαδικασίες της Επιτροπής Μεταφορών. Μπορώ λοιπόν να πω ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει πραγματικά να παρουσιάσουμε ένα αντίβαρο όσον αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό ε, των οποίων ε, αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι η συνεβαστική λύση θα μπορούσε να είχε διευρυνθεί. Κρίμα που δεν έγινε, αλλά ε, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν διαφορετικές ταξινομήσεις και διαφορετικές κατηγορίες. Αύριο πρέπει να ψηφίσουμε. Θετικά, θετικά, για να επιβεβαιώσουμε τη θέση μα. Η Επιτροπή Μεταφορών αναμένει ακριβώς αυτή την απόφασή μας και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Τόμας Μαν για την εξαιρετική εργασία που έκανε και τις έντονες προσπάθειες του να επιτύχει μια συμβαστική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε, κυρία Χίρσ θέλω και εγώ να μιλήσω ως ομάδα των ε, πολιτικών ελευθεριών είχαμε απορρίψει τότε την πρόταση και πάλι θα το κάνουμε, θα απορρίψουμε διότι πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανισορροπία. Βεβαίως εδώ θέλουμε να προσπίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών. Δεν είναι δυνατόν συνέχεια να τους φέρουμε σε πολεμικές, σε πολεμικές συγκρούσεις. Τι δύο αυτές πλευρές. Διότι αν φυγούν, αν υποφέρουν ας πούμε οι εργοδότες θα χαθούν σε εργασίε του εργαζόμενο. Λοιπόν, πιστεύω ότι εδώ γίνεται υπερβολική απλούστευση και εάν ε, γίνει αλλαγή θα υπάρχουν πολύ μεγάλοι, θα, ε, θα επιβληθούν πολύ μεγάλοι περιορισμοί. Εκτός τούτου, αυτή η ποιοτική πτυχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας συνεχούς ε, κατάρτισης ε, την οποία θα δεχτούν οι εργαζόμενοι, θα δεχτούν να συμμετάσχουν. Αλλά δυστυχώς αυτό το θέμα της ε, κατάρτισης και αυτό απορρίφθηκε και γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους που καταψηφίσαμε. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Χέντελ. Χέντελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μια σύντομη παρατήρηση. Ούτε και εγώ καίγομαι να υπεραμυνθώ του συμβιβασμού που επιτύχαμε. Ήθελα ε, κάτι πολύ σαφέστερο και καλύτερο. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε όλη αυτή τη ε, συζήτηση στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή Μεταφορών περιμένει. Τώρα, αυτό που είναι σαφές μεταξύ των δύο επιτροπών είναι το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης. Ιδίω το θέμα των υπεργολαβιών. Εκεί υπάρχουν θαυμάσιες ε, προτάσεις, διότι οι υπεργολαβίες και όλο αυτό το ζήτημα των υπεργολαβιών κινδυνεύει να γίνει ένα τεράστιο dumping προς όφελος της χαμηλής και κακής ποιότητας. Από ό,τι ξέρω εγώ στην Επιτροπή Μεταφορών το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται με τεράστιες δυσκολίες. Γι' αυτό παρακαλώ τον συνόδελφο μου κύριο Μπαχ στην Επιτροπή Μεταφορών να κλείσει τέλος πάντων αυτή, αυτό το παρασυράκι και εμείς ε, θα καταψηφίσουμε όλες τις διαγραφές κοινωνικών κριτηρίων. Φαίνεται ότι η Επιτροπή Μεταφορών υπερασπίζει τις διαγραφές κοινωνικών κριτηρίων. Εμείς ε, εάν δεχτούμε μία, ένα no-go, δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να, να με κοινωνικά κριτήρια και την προάσπιση των κοινωνικών κριτηρίων. Έτσι θα, θα προσωπήσουμε τη θέση μας στο, στο, στην Ολομέλεια. Ο κύριος Μάν. Ευχαριστώ για την ε, διευκρίνηση. Είναι σαφές, όταν έχουμε συμβιβασμούς, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λίγη υποχώρηση από τη μία πλευρά, λίγο κέρδος από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό σας είπα, μπορούμε όλοι να συναντηθούμε στην, κοινή, γραμμή, στην κοινή βάση. Ακριβώς αύριο θέλουμε να επιβεβαιώσουμε αυτή τη θέση μας. Ε, Κα, ε, κανένας δεν θέλει να ε, υποστούν βλάβη οι εργαζόμενοι λόγω θέμη του ανταγωνισμού. Κανένας δεν θέλει κοινωνικό dumping, κανένας δεν θέλει επιχειρησιακές ε, απώλειες ε, και πρέπει να, εξετάσουμε και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό ακριβώς εγώ περιορίζουμε στο ρόλο, στο ρόλο μου ως εισηγητού. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα ως σκιώδης από την Επιτροπή Μεταφορών και τους κοιόδης της Επιτροπής Απασχόλησης να συναντηθούμε για να εξετάσουμε ακριβώς θέματα όπως οι υπεργολαβίες και μια άλλη σημαντική απόφαση που πρέπει να εξετάσουμε ένα, μια ρήτρα επικουρικότητας, δηλαδή αυτός ο ενδοκοινοτικός ανταγωνισμός, ενδοενωσιακός ανταγωνισμός. Εμείς θέλουμε και μία ανακοίνωση της Κομισιόν και όχι στοιχεία από τις Κομισιόν που να μας δυσκολέψουν περισσότερο το έργο. Ε, ε, ε, θα πρέπει να τα εγκρίνει αυτά η Κομισιόν και αυτό θα το συζητήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όμως ξέρω ότι οι εργαζόμενοι του τομέα αισθάνονται ότι υπάρχει μια δύναμη υποστήριξης ε, πίσω, πίσω τους ε, και ότι δεν τους έχουμε εγκαταλείψει. Εάν αύριο μπορούμε να επιτύχουμε μία υπερψήφιση, τότε το μήνυμα που θα δώσουμε είναι ήδη σημαντικό προς την Επιτροπή Μεταφορών. Μετά η Επιτροπή Μεταφορών θα κάνει τη δική της διαβούλευση και θα κάνουμε μια κοινή συνάντηση με τους κοιόδης ε, ε, μεταξύ απασχόλησης και μεταφορών ξέρουμε και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι ε, αυτό το οποίο επιζητούμε θα γίνει με κοινέ προσπάθειες. Δεν είναι ότι θα είναι μία επιτροπή αρμόδια και όλοι οι άλλοι ας πούμε απλώς ε, εκφράζουν την άποψή τους. Εμείς θέλουμε και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να υπάρχει ίση και δίκαιη μεταχείριση. Και ε, προς αυτό το στόχο οδεύουν όλες μας οι προσπάθειες. Ωραία, θα ψηφίσουμε αύριο ακριβώς τις υπηρεσίες εδάφους, στο θέμα 13. Ατζέντα για επαρκή ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν είναι συγγήτρια. 303 τροπολογίες για σήμερα. Ο λόγος του κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολλέ τροπολογίες, όπως είπατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε. Αλλά ευτυχώ υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, πολυάριθμε, που μπορούν να αποτελέσουν βάση για να συμπληρώσουμε τα όλα όσα έχουν υποθεί. Αλλά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όμως ορισμένα σημεία. Υπάρχει βέβαια υποστήριξη ευρεία ότι οι συντάξει του πρώτου πυλώνα είναι σημαντικές και αυτός ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να αποτελεί ε, το, το βασικό κομμάτι της σύνταξης. Υπάρχουν επίσης άλλες τροπολογίες για αυτό τον πρώτο πυλώνα φορολογικά κίνητρα πιο συγκεκριμένα. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που αφορούν τον αριθμό που έχει δουλέψει, των ετών που έχει δουλέψει κανείς, όχι την ηλικία συνταξιοδότησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τους δύο παράγοντες. Ε, υπάρχει μια υποστήριξη για το 121 και 122 για τις συντάξεις του πρώτου πυλώνα. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα. Όταν εξετάζω τις τροπολογίες που όπως η 44, 68, 69 και η 71, ε, αυ, με αυτές τις τροπολογίες δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι όχι μόνο ο πρώτος πυλώνας, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι σημαντική, υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά. Και είμαι κατάπληκτη με τις τροπολογίες ε, των πράσινων. δηλαδή που λένε ότι το σύστημα των πολλαπλών πυλώνων δεν είναι θετικό. 103, 117 και 118. Δεν συμφωνώ με αυτές. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα με αυτές τις τροπολογίες, οι οποίες δεν επιθυμούν να υπάρχει σχέση ανάμεσα στο προσδόκιμο ζωής που είναι μεγαλύτερο σήμερα και στην ηλικία ταξιοδότησης ε, θεωρούν ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Επίση υπάρχουν ανθρωπολογίε που λένε ότι τα συστήματα υγεία με βάση τα οποία έχουμε αποταμιεύσει ε, είναι υποπίεση. Μεγαλύτερη πίεση μάλιστα από τα συστήματα τα pay as you go. Συμφωνώ με αυτή την ιδέα. Αλλά δεν συμφωνώ με την τροπολογία 150 που περιορίζει την ε, ελευθερία κεφαλαίων για τα συνταξιδοτικά ταμεία. Την ελευθερία δηλαδή διακίνηση των κεφαλαίων. Είμαι πεπισμένη, κυρία Πρόεδρε, ότι η ενισχυμένη συμμετοχή των ε, εργαζομένων είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που μπορεί να μας εξασφαλίσει μια επαρκή βάση, ούτω ώστε να έχουμε μια σύνταξη πρώτου πυλώνα, η οποία εγγυάται ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Αξιοπρεπές εισόδημα από τον πρώτο πυλώνα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει περισσότερα άτομα να είναι στην αγορά εργασία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά και όλα τα μέτρα ε, δυνάμει των οποίων τα άτομα άνω των 50 που θέλουν ακόμα να εργαστούν να μπορούν να το κάνουν. Βλέπω χώρες όπως το Βέλγιο, 5% άνω των 60 είναι ενεργοί. Δεν είναι δυνατόν όμως αν έχουν προσδόκιμο ζωής 80 χρόνια. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματική ηλικία, αλλά συμφωνώ από την άλλη ότι πρέπει να εργάζονται, να είναι ενεργά περισσότερα άτομα. Με αυτό ακριβώ το πνεύμα νομίζω ότι μπορώ να βασιστώ στην υποστήριξη των σοσιαλιστών. Το θετικό, ε, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι υπάρχουν και πολλές τροπολογίες για τις γυναίκες. 229, 230, 234, 238. Για την 150, 180, 270. Αυτές αφορούν ε, την πολύχρονη εργασία. Υπάρχουν και καλές προσθήκες για τους ε, ανθρώπους που έχουμε λίγο εγκαταλείψει τους μακροχρόνια άντρους κτλ. και που θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή εργασία. Επίσης υπάρχουν και τα ευπαθή άτομα, υπάρχουν παρατηρήσεις που τα αφορούν, που όλο να δεχτώ αυτές τις παρατηρήσεις για τα ευπαθή άτομα και τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αν πρέπει να πούμε, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να δουλέψουμε περισσότερα χρόνια, αυτό το, αυτή την απόφαση δεν την παίρνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών, σε Διαπραγματεύσει με του κοινωνικού εταίρου. Θα ήθελα να, κάνω κάποιες, να δώσω κάποιε διευκρινήσει για αυτό το σημείο. Εκεί που έχω μεγάλα προβλήματα είναι η διαγραφή της παραγράφου 8, ε, η τροπολογία 176 των πράσινων που αφορά αποκλειστικά τον πρώτο πυλώνα. Όταν υπάρχει πρόβλημα με τα δημόσια οικονομικά, το πρώτο πράγμα που περικόπτουμε είναι οι συντάξεις. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, τι κάνανε. Αυτό ακριβώ. Αν κανένα δεν αποταμίευσε για τη σύνταξή του και αν εξαρτάται από την κυβέρνηση και την κρατική σύνταξη, το πρώτο πράγμα που περικόπτεται όταν έχουμε δυσκολίες όπως διαπιστώσαμε είναι ακριβώς αυτό. Το 2020 θέλουμε να έχουμε αξιοπρεπές εισόδημα από το πρώτο πυλώνα. Γι' αυτό ακριβώς, αν θέλουμε κάτι τέτοιο, χρειάζονται διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, διαρθωτικές αλλαγές. Αν ε, κλείσουμε τα πράγματα στη δημογραφική πραγματικότητα, θα έχουμε προβλήματα. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την εθελοτυφλία. Θα πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένε, εγγυημένε συντάξει, αλλά δεν μπορούμε απλώ να τα αναπούμε. Ναι, θα αυξήσουμε τα πριμ ή θα προσπαθήσουμε να, δούμε, να βρούμε άλλα ε, οικονομικά μέσα για να εξασφαλίσουμε τη συντάξη. Γιατί αν κάνουμε κάτι τέτοιο, αυτό θα γίνει εις βάρος κάποιων άλλων υποθέσεων, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υποθέσεων, του κράτους πρόνοια κτλ. Γι' αυτό ακριβώς, Πρόεδρε, θα πρέπει όλοι μαζί να δείξουμε επικοδομητικό πνεύμα, συνεργασία και στα πλαίσια της ιδέας της αλληλεγγύης μεταξύ των γενναίων να μην πιέσουμε απόλυτα μέχρι να τους συνθλίψουμε τους νέους οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν ένα πολυάριθμο, ας πούμε, μια πολυάριθμη κατηγορία ηλικιωμένων σε αυτά τα πλαίσια δηλαδή αυτού του πρώτου πυλώνα θα, θα την πληρώσουν οι νέοι για αυτή την πολυάριθμη ομάδα ηλικιωμένων. Θα πρέπει να βρούμε και άλλα μέσα χρηματοδότηση. αλλά και αυτά τα μέσα δεν είναι ανεξάντλητα, μην νομίζετε, ούτε απεριόριστα. Γιατί ε, όταν ξοδέψουμε τα λεφτά, τελειώσανε μετά. Για τα, από τα υψηλότερα εισοδήματα πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη ε, αλληλεγγύη, φυσικά. Αλλά δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο μόνο να εξαλείψουμε την πίεση. Δεν θέλω να επιβάλλω συμπληρωματικέ συντάξει, επικουρικέ συντάξει κτλ. Και φοβάμαι ότι είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν αυτή τη δυνατότητα με ένα πολύ προσεκτικό τρόπο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διάφορες γενιέ επίσης να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και να το σκεφτούν μαζί το θέμα. Για τον πρώτο πυλώνα όλες οι ιδέες Κάποιες ιδέες υποστηρίζω. Ε, θέλω να υπάρχουν πληροφορίες για τις ε, συντάξεις και οι τροπολογίες που μιλάω για τις πληροφορίες για τις συντάξεις υποστηρίζω και όταν μιλάμε για το δεύτερο πυλώνα μιλάμε για την υποχρεωτικότητά του. Δεν έχει νόημα να έχουμε ένα δεύτερο πυλώνα. Αν υπάρχει όμως τα πλαίσια της αλληλεγγύης ε, ένας δεύτερος πυλώνας, τότε θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Υποχρεωτική συμμετοχή λοιπόν στο δεύτερο πυλώνα. Αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση να έχουμε ντε και καλά ένα δεύτερο πυλώνα. Αν υπάρχει όμως υποχρεωτική συμμετοχή. Ορισμένοι συνάδελφοι μου ψιθυρίζουν διάφορα. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση, ας πούμε. Να μην έχουμε υποχρεωτικά ε, δεύτερο πυλώνα. Αν όμως έχουμε, τότε θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής αυτών. Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε επίσης ότι υπάρχουν τόσο, μικρομεσές, τόσο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υποχρεωθούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα σύνταξη δικό τους. Υπάρχουν όμως δημιουργικές ιδέες. Ας πούμε, όταν έχουμε μία μικρή επιχείρηση, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν παραδείγματα. Θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη για τις δυνατότητε αυτές για τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν συμφωνώ με τις τροπολογίες που καταργούν 140, 141, 145 που θέλουν να καταργήσουν ή να αποδυναμώσουν το δεύτερο πυλώνα. Και δεν θέλω επίσης να μειώσουμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Εγώ το σκέφτηκα αυτό το θέμα. Σκέφτηκα ότι ίσως ε, αυτή η αλληλεγγύη για να την διατηρήσουμε θα πρέπει να εντάσσεται και στον δεύτερο πυλώνα. Ε, πρέπει εκεί να μιλήσουμε για τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και για τις διάφορες γενιές οι οποίες εμπλέκονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει και ένα πρόβλημα για την 253 και 254 τροπολογία. Όντω χρειάζονται περισσότεροι κανόνε για την προστασία των συνταξιδοτικών ταμείων, των ιδιωτικών συνταξιδοτικών ταμείων. Φρέντερικ, η τροπολογία σου για το care credit. Ναι, είναι μια δυνατότητα αυτή. Τα άτομα δηλαδή τα οποία α, έχουν κάποια, κάποια θεραπεία κτλ. να παίρνουν και τη σύνταξή τους παρόλα αυτά. Επίσης για τους μετακινούμενους ε, εργαζόμενους. Το Συμβούλιο ξέρουμε ότι ασχολείται να προσπαθεί να προετοιμάσει μια κοινή θέση μετά από την έκθεση της οποίας ήμουνα εισηγήτρια. Αλλά δεν έχει ακόμα καταλήξει το θέμα. Εμείς ως Κοινοβούλιο είπαμε ότι η μεταφορά των συντάξεων πρέπει να υπάρχει. Το τα δικαιώματα τα οποία έχουμε συσσωρεύσει σε ένα άλλο συνταξιοδοτικό ταμείο, σε ένα άλλο κρατος μπορούν να διατηρηθούν και μπορούν να εξελιχθούν σύν το χρόνο. Υπάρχει αυτή λοιπόν η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών. Μερικές φορές όμως δημιουργούνται προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε ε, μεταφορά των κεφαλαίων αν οι άλλες συνθήκες υπάρχουν. Είπα στους πράσιους ότι αν σε μια χώρα δεν αμφισβητείται η μεταφορά, είδα ότι μετά από τις αλλαγές στα συστήματα δεν, μπορούμε να, δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το κεφάλαιο, να εγγυηθούμε το κεφάλαιο, απλώς να εγγυηθούμε τα δικαιώματα. Αυτό το, αυτή όμως την ιδέα την απορρίπτω. Υπάρχει και ένα πρόβλημα με τον Τόμας. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο και εδώ συνεχίζεται η διαπραγμάτευση να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για την δημιουργία συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Εγώ, εσύ δεν συμφωνείς, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έτσι. Γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτήν την περίπτωση μεταφορές. Αν πούμε, από τα 21 χρόνια, ας πούμε, ή 23 χρόνια, αρχίζουμε να δημιουργούμε το συνταξιδοτικό μας δικαίωμα, Και υπαρχουν κάτι κράτη-μέλη που λένε ότι ανεξάρτητα από την ηλικία, ε, από τη στιγμή που αρχίζουμε να εργαζόμαστε, ε, δίνουμε εισφορέ για τη σύνταξη. Αν όμως ε, μετά από τρει μήνε φύγουμε από αυτή τη χώρα και πάμε σε μια άλλη επιχείρηση, α πούμε, πρέπει να κρατήσουμε αυτού τους τρεις μήνες. <laughs> Αυτό τότε τι δημιουργεί, δημιουργεί τεράστιο διοικητικό χάος. Μακριά από εμά. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο για την δημιουργία σταξιδιωτικού δικαιώματος το να προβλέψουμε αντί μια κάποια περίοδο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, ας πούμε, ε, η περίοδος είναι πέντε χρόνια. Ε, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την κινητικότητα των εργαζομένων και την παράλληλη μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Κοιτάξτε κυρία Πρόεδρε τι θα κάνω. Θα προσπαθήσω να προετοιμάσω ένα κείμενο και θα συμπεριλάβω κάποιες τροπολογίες Εν συνεχεία, θα γίνει μια διαβούλευση. Θα προσπαθήσω να δω ποια είναι η θέση μας συνολικά. Υπάρχουν, τόσα, υπάρχουν κάποια πολύ αμφισβητούμενα σημεία και δεν θέλω να επιβάλλω τις δικές μου ιδέες, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν σημεία που μπορούμε να συμφωνήσουμε και αυτά θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω στο κείμενο. Την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε μια συνεδρίαση με τους σκιώδεις συζητητές, προβλέπετε αυτό. Και εκείνη τη μέρα η κόρη μου θα πάρει το διπλωμά της. Το πρόβλημα είναι ε, ότι εγώ θέλω να πάω σε αυτή την ε, τελετή. Ε, θέλω λοιπόν να αλλάξετε την ημερομηνία ε, συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση, γιατί η συντάξη είναι κάτι τόσο πολύ σημαντικό για την ευημερία μα για το βιωτικό μα επίπεδο. Για πάρα πολλά άτομα είναι σημαντικό αυτό το θέμα, όλο και περισσότερα. Έτσι. Γιατί το 1 πέμπτο του πληθυσμού μα είναι μεγαλύτερο από 50 χρόνια. Είναι μια κάποια ηλικία και επομένω είναι και η ώρα να δράσουμε. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να ζήσει πολλά χρόνια, ευτυχής, σε καλή υγεία, αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται και λεφτά και επαρκές εισόδημα. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την τοποθέτηση. Ο λόγο τους και οδησηγητές. Επτά μέλη συγκεκριμένα που θέλουν να λάβουν το λόγο. Στις 11.30 όμως πρέπει να ξεκινήσουμε την ακρόαση. Παρακαλώ Δύο λεπτά ο καθένας το πολύ. Ο Νταρντά. Merci, Madame la Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και η συγγήτρια, είναι πολύ άριθμες οι τροπολογίες. Και εγώ μόνο πάνω από 50 υπέβαλα. Έχω συνεισφέρει πολύ λοιπόν σε, αυτή την, σε αυτόν τον πολλαπλασιασμό. Ε, Θέλω απλώ να συμβάλλω στη βελτίωση του κειμένου. Ε, οι τροπολογίες μου ε, μάλλον ε, συστιάζουν συγκεκριμένα θέματα, κυρίως δύο θα σχολιάσω εγώ. Το ένα είναι το θέμα της, ε, του μίξ των ε, πυλώνων και το νομικό θέμα των, ε, της, των συνταξεών. και πιο συγκεκριμένα της ηλικίας συνταξιοδότησης. Ε, ο πρώτος πυλώνας είναι ε, θεμελιώδης. Είναι ο πυλώνας που δίνει τη μεγαλύτερη ασφάλεια, που είναι ο πιο αλληλέγγυος. Η συνταξιοδότηση πρώτη πυλώνα δεν θα πρέπει να είναι η ελάχιστη, θα πρέπει να είναι ένα εισόδημα ε, που θα υποκαθιστά τον μισθό σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα, προτεραιότητα είναι η απασχόληση. Όσο πιο πολύ απασχολούνται, τόσο πιο εύκολο να χρηματοδοτηθεί ο πρώτο πυλώνα. Επίση θα πρέπει να σκεφτούμε και εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότηση. Μια γενικευμένη, για παράδειγμα, ε, κοινωνική εισφορά. Ο πρώτο πυλώνα, βέβαια θα πρέπει να συμπληρώνεται από ένα δεύτερο πυλώνα, πιστεύει η ομάδα μα τουλάχιστον. Ε, ένα συμπληρωματικό γενικό ε, οριζόντιο πυλώνα που θα τον διαχειριζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους που θα επενδύουν σε αυτό το πυλώνα με βιώσιμο τρόπο και οι ε, εργοδότες θα αναλαμβάνουν και αυτή ευθύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεπερνάω το χρόνο, αλλά είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Οπότε, σε σχέση με αυτό το, σε αυτούς τους πυλώνες, επηρεάζεται ο καθένα από το σύστημα της χώρας στην οποία ζούμε. Είναι προφανές. Και κάθε ένα από αυτά τα συστήματα έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. θα πρέπει να βασιστούμε στις γενικές τάσεις, ε, ε, να λάβουμε υπόψη την επικουρικότητα και να υποβάλουμε προτάσεις που να μπορούν να εφαρμοστούν παντού. Όχι να μεταγράφουμε για, σε όλους το σύστημα μιας χώρας. Παρόλο ότι ένα σύστημα που να λειτουργεί μια χαρά σε μια χώρα, για παράδειγμα το σύστημα των κάτω χωρών, όμω αυτό δεν το κάνει ιδανικό για τι υπόλοιπε χώρε. Σε ό,τι αφορά το θέμα τη ηλικία δεξιοδότησης. Ε, συγγνώμη, θα, θέλατε να παραμείνετε να περιουστείτε στα δύο λεπτά τα οποία σας δώσαμε. Έχετε ξεπεράσει τα τρία λεπτά ήδη. Πολύ λίγο έχω ακόμα. Ε, δεν θα πρέπει να είναι αυτή η προτεραιότητα. Θα έπρεπε να εργαστούμε καταρχήν στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότηση και στον αυτό. Ε, στην αυτόματη εξέλιξη της ηλικίας δεξιοδότησης, της ε, κατανόμων ηλικίας δεξιοδότησης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έτη ε, ε, φορών, ε, το δίκτυο ενεργείας κλπ. Ευχαριστώ ο κύριος Ντεμπάκερ και μετά κύριος Χέντελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω υποβάλει πολλέ τροπολογίε. δεν σα εκπλήττει όμω το γεγονός ότι εμείς περισσότερο συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Υπάρχει μία δέσμη κρατών ε, μελών ε, που έχει αντιρρήσεις, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε και έναν τρίτο πυλώνα για την αηφορία. Είναι απολύτως απαραίτητο. Ορισμένοι πιστεύουν ότι μόνοι, ο πρώτος πιλότας επαρκεί. Αυτό είναι σαφώς λάθος. Θα πρέπει να δούμε και το ιστορικό παρελθόν, πώς εξελίχθηκαν οι συντάξεις στην Ευρώπη, πώς πιέζονται τώρα λόγω των συνθήκων χαίρομαι για τις διαφαινόμενες λύσεις που υπάρχουν στο τραπέζι. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια αντίληψη της πραγματικότητας μεταξύ των γενεών και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία στο μέλλον ε, θα τα εφαρμόσουν ε, οι επόμενες γενιές. Ίσως μέτρα λοιπόν τα οποία δεν τολμούμε να τα λάβουμε σήμερα, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να ληφθούν. Θέλουμε επίσης να υπάρχει αυτό το θέμα ανείχνευσης για τα διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Πρέπει να είναι απόλυτα ε, διαφανής η διαδικασία δημιουργίας των συντάξεων για τους πολίτες. Εν συντομία, Όσον αφορά το πλαίσιο, υπάρχουν ήδη κανονιστικές ρυθμίσεις για τον ασφαλιστικό τομέα, όμως χρειάζομαστε και το στοιχείο της ελαστικότητας για να μπορούν τα συστήματα αυτά, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο, να καλυφθούν. Τέλος, θα πρέπει να αυξηθούν, ε, αυξηθεί η συνταξιωτική ηλικία. Η ηλικία λοιπόν που θα παίρνει κάποιος τη σύνταξη δεν μπορεί να είναι 60. Τώρα ζει ο κόσμος μια χαρά μέχρι το 85 και δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια να καταβάλλονται συντάξεις. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί το όριο. Αν θέλουμε αηφορία στις συντάξεις θα γίνει και αυτό. Ο Χέντελ και μετά η κυρία Ρεγκίνα Μπάστος. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ επειδή μας πιέζει ο χρόνος θα είμαι σύντομος. Ε, εμείς έχουμε κάπως παρεκκλίνουσα άποψη από το κύριο ρεύμα ε, εδώ εμπλέκονται ε, δημοκρατικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία και που σαφώς επηρεάζουν ε, τα, τις τελευταίες δεκαετίες τα κράτη-μέλη. δεν συμφωνούμε παρόλο και αν υπάρχει το σενάριο της χειρότερης κρίσης θα επέλθει μια τέτοια οικονομική ανάπτυξη και αύξηση ώστε μέχρι το 2030 θα έχει αναστραφεί τελείως το κλίμα και θα μπορούσαμε να υπάρχει, να έχουμε ένα ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτήσει πολύ ωραίες και ικανοποιητικές συντάξεις για τους ηλικιωμένους. Πρέπει να ε, επαναέλθουμε ε, σε μια ισότιμη χρηματοδότηση και κάλυψη των ε, συντάξεων. Ε, δεν μπορούμε εδώ να έχουμε μία διαφοροποίηση των συντάξεων βάσει του ταμείου στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος. Πρέπει να δούμε κάθε εργαζόμενος τι έχει προσφέρει στην εταιρεία έτσι ώστε να έχει ισότιμα δικαιώματα με τους άλλους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική ε, η οποία να είναι δίκαιη και θεμητή δεδομένου ότι ο κατώτερος μισθός, τα εισοδήματα μειώνονται συνέχεια. Δεν έχουμε αντίρρηση στην ε, βελτίωση της, ε, των εισφορών της βάσης εισφορών. Αλλά θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η προστασία των αδυνάμων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στην ε, κεφαλουχική αγορά, στήριξη της, του πρώτου πυλώνα, ενίσχυση του πρώτου πυλώνα, πρέπει να επανέλθουμε στην αηφόρο ανάπτυξη ρητός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάστος και μετά ο κύριος Μπεκέα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Καταρχήν συγχαίρω ε, την ε, Ρία για την έκθεση της αυτή. Ήμουν ε, ε, εισηγείται εκ μέρους της ομάδας ε, γυναικών, της Επιτροπής Γυναικών. Ε, έχουμε δύο βασικά ζητήματα εδώ. Τη γύρανση του πληθυσμού, που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των συνταξιωτικών συστημάτων σε όλες τις χώρες μας, ιδιαίτερα στις χώρες που πλήττονται αυτή τη στιγμή από σοβαρές οικονομικές χρηματοοικονομίες και Κοινωνικέ ε, κοινωνικές κρίσεις όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Δεύτερο, ε, ένα, μέρο, ένα σημαντικό μέτρο ε, είναι η δάνεια, πιστώσεις προς άτομα τα οποία έχουν υπό τη φροντίδα τους άλλα άτομα τα οποία εξαρτώνται από αυτά. Είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο προβλέπει σε ορισμένα κράτη-μέλη και συμφωνώ με τις ιδέες της εισηγήτριας για πολύ επικαιρά θέματα όπως η ανάγκη να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής η ηλικία στην αξιοδότηση, όπως επίσης και η ε, μάθηση, διαβίου μάθηση, η, ο συνδυασμός ε, προσωπικής επαγγελματικής ζωής και ε, οι προβλέψεις για γύρανση του πληθυσμού. Κάτι που θα έπρεπε να υπογραμμιστεί και το καθιστά σαφές η συγκήτρια είναι η ε, η ε, συνταξιοδότηση των ε, γυναικών και των νέων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δείτε ευκαιρία στους, στους τους εργαζόμενους που θα συνταξιοδοτηθούν ε, να συνεισφέρουν περιοδικά ε, και τακτικά για τη σύνταξή τους έτσι ώστε να αυξηθεί αυτή ε, όταν συνταξιοδοτηθούν. Μία ακόμα φορά θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Μπεκέρ, ο Ρίμαν, Μακεντάιρ και εκεί τελειώνουμε. Ο κ. Μπεκέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Έχουμε εδώ μια έκθεση. η οποία αφορά όχι μόνο το εν τρίτον του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά και τη χρονική, το χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2060. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη καινούργια γενιά που θα συνταξιοδοτηθεί. Έχουμε λοιπόν μια ευθύνη για όλους τους Ευρωπαίους και δεν έχουμε αρκετό χρόνο σε αυτή την Επιτροπή να συζητήσουμε ενδελοχώς το ζήτημα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να κάνουμε μία εις βάθος συζήτηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω επί της ουσίας, αλλά εδώ πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και πρέπει όλα τα κράτη-μέλη και όλοι οι υπεύθυνοι να συμφωνήσουν προφανώς να στηρίξουν τον πρώτο πυλώνα, να διαμορφώσουν ε, με ρεαλισμό το δεύτερο πυλώνα και με όλες τους τις δυνάμεις να φροντίσουν για μία σωστή και αξιοπρεπή... Ε, α, να διαγραφούν οι όροι ελάχιστη σύνταξη. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ε, εξασφάλιση μιας βέλτιστης ζωής. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε κάτι, να αποφασίσουμε ε, κάτι το οποίο θα ε, βλάψει ε, το, το όριο αξιο, αξιοπρεπούς διαβίωσης εκατομμυρίων Ευρωπαίων τώρα και στο μέλλον. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό στο μέλλον. Ο κ. Σωρή και μετά ο κύριος Τομασμάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. 27 κράτη-μέλη με 27 διαφορετικά συνταξιδοτικά συστήματα, διαφορετικές παραδόσεις. Οπότε το θέμα δεν είναι ένα θέμα διαλόγου μεταξύ πολιτικών ομάδων μόνο. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω το σημείο 4 του κειμένου, παράγραφο 4, όπου η Ρία υπογραμμίζει υπογραμμίζεται υπάρχει δι, ε, κρίση κλπ. Όλα αυτά. Μιλά για το συνταξιωτικό σύστημα που έχει διάφορους πυλώνες και εδώ συμφωνώ και μετά μας δίνει παραδείγματα. Δημοκρατικό πυλώνας με μια αξιοπρεπή ελάχιστη σύνταξη, ε, δεύτερος ε, πυλώνας με συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων και τρίτος πυλώνας που είναι ιδιωτική ασφάλιση. Όλα αυτά πολύ καλά. Αυτό που δεν με βρίσκει σύμφωνο είναι το μοντέλο το μοντέλο που θέλει να προτείνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε τους ορισμούς. Ο ορισμός ο ίδιος αγνοεί το γεγονό ότι ορισμένες χώρες μπορούν να χρησιμοποιούν το μοντέλο benchmark. Ο πρώτος πυλώνας για ορισμένες χώρες δεν είναι ελάχιστη σύνταξη. Σε ένα τέτοιο σύστημα ε, ο ρόλος του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα αλλάζει. Μπορεί να υπάρχει σύστημα ε, με ένα βασικό πυλώνα. Συνεπώς ε, δεν είναι δυνατόν να ε, θεωρήσουμε ότι ο δεύτερος πυλώνας θα είναι υποχρεωτικός. Λέγοντας κάτι τέτοιο αγνοείται το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Ένα λεπτό και 47 δευτερόλεπτα. Ωραία, άρα έχω, μου περισσεύει λίγος χρόνος. Έχω υποβάλει τροπολογίες για αυτό το θέμα. Ε, είμαι και πάλι υπέρ της διάδοση του, της μεθόδου του δεύτερου πυλώνα, αλλά όχι να είναι υποχρεωτικός. Ευχαριστώ ο κύριος Τόμας Μαν, ε, εισηγητή Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Με ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος ε, ο Σενάλφος Μπέκερ. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο δεδομένου ότι εδώ αφορά όχι μόνο εκατομμύρια του πληθυσμού μας αλλά και γενιές. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους νέους, ε, τη νέα γενιά και τις καινούργιες, τις επερχόμενες γενιές τελείως απροστάτευτες. Χρειάζεται θεσμικά να τις προστατεύσουμε και να τους πούμε ότι θα υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Ε, η Ρία εκπώνησε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Εγώ είμαι εισηγητή στην Οικονομική Επιτροπή και με την Επιτροπή Απασχόλησης έχουμε βεβαίως μαζί αρμοδιότητες αλλά έχουμε και άλλες αποκλειστικέ αρμοδιότητες. Εχθέ στην ε, συνάντηση των σκιωδών ε, καταφέραμε μια μεγάλη συμφωνία, α πούμε, ευρεία συμφωνία. Και ελπίζω ότι ακόμα και εδώ ε, στις, στα, στις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσώπων των εργαζαμένων του σώματος ε, αφορούν όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Έχουμε πει ότι και οι δύο πυλώνες πρέπει να παραμείνουν δεν μπορούμε να τις φέρουμε σε αντίθεση και οι δύο έχουν το ρόλο να παίξουν, δεν πρέπει να τις αποδυναμώσουμε με κανένα τρόπο. Έχουμε, έχω εξετάσει μεγάλη τεκμηρίωση ε, για συνταξιδετικών θεμάτων από τα κράτη-μέλη. Εμείς συμφωνούμε οι κοινωνικοί εταίροι να ε, ε, εμπλακούν, να, να συμμετάσχουν και να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε διαφορετικές γενιές, όχι μόνο στους συνταξιούχους ή στους προσυνταξιοδότηση. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο μία ηλικιακή ομάδα, αλλά πολλές. Παρακαλώ λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα αυτό ε, με, σοβαρότητα, εις βάθος και ενδελεχώς και ευρύτατα. Δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι στο γόνατο. Πιστεύω ότι έχουμε επαρκή χρόνο για να, για να το εξετάσουμε εις βάθος. Η κυρία Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Όπως είπαν και οι άλλοι, αυτό το, αυτός το φάκελος είναι εξαιρετικά επίκαιρος και σημαντικός και εγώ συμφωνώ με την ε, παράκληση να έχουμε περισσότερο χρόνο προς συζήτηση. μεγαλύτερη μου επιφύλαξη είναι να έχουμε ε, μία λύση η οποία να καλύπτει τα πάντα. Δηλαδή ε, ένα, ένα κουστούμι κομμένο και ραμμένο στις διαστάσεις όλων. Ορισμένα προγράμματα χρειάζονται ριζική ε, αναθεώρηση, αλλά δεν θέλουμε ε, λόγω βιασύνης να επιφέρουμε ζημιές ή τις οποίες απρόσκοπτες, δεν είχαμε υπολογίσει. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις όσον αφορά τον πυλώνα. Σε ποιο πυλώνα ανήκει η εργασία για το συνταξιδοτικό πλαίσιο, στο 1 ή στο 2. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πυλώνα 3 για την ε, για το στοιχείο της μεταφοράς των συντάξεων, την κινητικότητα των συντάξεων. Εγώ θα συμμετάσχω πλήρως ε, στις ε, συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια Μιλήσατε ήδη 15 λεπτά στην εισαγωγή, Δύο λεπτά τώρα σας περισσεύουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τον πρώτο πυλώνα. Του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ε, κι εγώ το ίδιο. Ε, οι συντάξεις είναι οι πρώτες οι οποίες ε, πλήττονται όταν πέφτουμε σε οικονομική κρίση. Οπότε, αν θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση στον πρώτο πυλώνα, δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε τίποτα γιατί είναι εθνική αρμοδιότητα. Αν τα κράτη-μέλη δεν το κάνουν, αυτό οφείλεται στο ότι δεν μπορούν και εμεί δεν έχουμε μέσα, μέσω του προπολογισμού μα, να κάνουμε τίποτε. Ε, υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, οπότε θα πρέπει να αρχίζουμε να αποταμιεύουμε για τη σύνταξή μας από ε, έτσι ώστε οι νέοι οι σημερινοί νέοι ε, να μην χρειάζεται ε, να στηρίζουν ε, τον γυράσκοντα πληθυσμό αργότερα. Συνεπώς, βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο, αλλά δεν αυξάνονται οι συντάξεις. Αυτό είπε ο συνάδελφός μας. Σωστό, έτσι είναι. Διότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι βιώσιμο να αυξάνονται οι συντάξει με τον προπολογισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο πρώτο πυλώνα είναι σημαντικό, αλλά είναι ουτοπικό να νομίζουμε, να φανταζόμαστε ότι όλα μπορούν να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα. Δεν επιβάλλω τίποτε, αλλά πιστεύω θα πρέπει να το σκεφτούμε. Και να πω και στον κύριο Σάμπα ότι ο τρίτος πυλώνας αφορά το άτομο. Εκεί δεν τίθεται θέμα αλληλεγγύης. Και δεδομένου δεν υπάρχει αλληλεγγύη, κάθε άτομο, κάθε εργαζόμενος μπορεί να ε, αποταμιεύει όσο θέλει. Γι' αυτό το λόγο και δεν είναι πρώτη μου επιλογή. Δεν μπορεί να είναι συμπληρωματική αυτή η σύνταξη. Ε, Πρόεδρος, ε, κάποιοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του. Ε, το κείμενο αυτό το συζητούμε περισσότερο από ένα χρόνο. Ο κ. Τομασμάν ζητάει περισσότερο χρόνο να του υπενθυμίσω ότι ε, καθυστερήσαμε τόσο πολύ έτσι ώστε η Επιτροπή ΕΚΟΝ να έχει χρόνο να το σκεφτεί. Την περιμέναμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Και στις 20 Μαρτίου θα δούμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Αν δεν είναι δυνατόν να το τελειώσουμε στην ώρα του, θα το ξαναδούμε. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Για το σημείο 15 δυστυχώς δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Ευχαριστώ την κυρία Μάκιντάιρ που δέχεται να το συζητήσουμε μετά την αημόσια κρόση. Περνάμε στο σημείο 17. Ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονές μας ε, που είναι ήδη μαζί μας και που άκουσαν το τέλος της προηγούμενης ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησης που αφορά επίσης τους ε, ε, εργαζόμενους που εργάζονται εκτός της χώρας τους. Η ακρόση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γνωμοδότης πρωτοβουλίας του κύριου Τόμας Χέντελ, όχι Τόμας Μαν που συνηθίζω να λέω, για τις διασυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον διεθνικό κοινωνικό διάλογο. Πριν δώσω το λόγο στους ε, τέσσερις προσκαλεσμένους μας, θα επιτρέψω εν συντομία στον κύριο Σιγητή να, όχι να μας παρουσιάσει την έκθεσή του βέβαια, αλλά να, να πει στους εμπειρογνώμονες τι περιμένει από αυτούς για να τροφοδοτήσουν και να εμπλουτίσουν τη συζήτησή μα, Ο κ. Συγητή. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Χέντελ. Τα ονόματα εντάξει, εδώ υπάρχει πάντοτε μια δοκιμασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οργανώνουμε αυτό την ακρόση, διότι εδώ πρόκειται για ένα πάρα πολύ περίπλοκο και δύσκολο θέμα που αφορά βεβαίως ε, τις ε, κοινωνικές ε, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Υπάρχουν προηγούμενα, ο, η έκθεση Alice, 2006 και Anderson 2008. Ε, εν τω μεταξύ βεβαίως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, έχουν προχωρήσει. Παραδείγματο χάρη το καθεστώς ε, του κοινωνικού διαλόγου. Αυτό έχει βελτιωθεί, έχει αναπτυχθεί, έχει ανέβει ψηλότερα. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, σχέσεις, επιχειρησιακές σχέσεις του τομέα των επιχειρήσεων δηλαδή. Έχουν και αυτές εξελιχθεί όσον αφορά τις επιπτώσεις των επιχειρησιακών συμβουλίων, εργασιακών συμβουλίων μέσα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, ο ρόλος τους είναι πιο έντονος από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Επίσης έχουμε περισσότερα πρωτόκολλα, μνημόνια και, ε, και δηλώσεις, δεσμευτικές δηλώσεις για διασυνοριακές ε, επιχειρησιακές δραστηριότητες. Έχουμε μια άλλη περιπλοκή, καινούρια, που και παραπέμπω από μια διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικές Πολιτικές Υποθέσεις ή μάλλον Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών Υποθέσεων. Ε, τρεις περιπτώσεις που ε, έκριναν την ε, κινητικότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων και το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τρεις περιπτώσεις λοιπόν της Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, εσωτερικών, εσωτερικών υποθέσεων, εσωτερικής διεύθυνσης, ε, πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, τις καινούργιες εξελίξεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το περιθώριο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις διασυνοριακές ε, σχέσεις, ε, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τους εμπειρογνώμονες να μας πούν τη γνώμη τους επ' αυτού. Έχουμε πολλά προβλήματα για αυτές τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον διάλογο. Πρώτον, κάθε κράτος μέλος έχει ένα τελείως άλλο σύστημα ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων. Ε, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε λοιπόν σε όλα αυτά τα περίπλοκα διαφορετικά συστήματα. Δεύτερον, τα κοινωνικά συστήματα στα κράτη-μέλη διαφέρουν πάρα πολύ και ε, Εμεί βεβαίω δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών μελών να διαμορφώνουν τι κοινωνικέ του συνθήκες. Αλλά ε, υπάρχουν πολλά κοινωνικά συστήματα που δεν λειτουργούν ικανοποιητικά και ε, υπάρχουν επιβαρύνσεις ει βάρο των εργαζομένων Γι' αυτό θέλουμε ακριβώς να επιτύχουμε τα ελάχιστα πρότυπα τα οποία είναι απαραίτητα για έναν σωστό ε, κοινωνικό ε, διάλογο και για, για δίκαιες συλλογικέ διαπραγματεύσεις και γι' αυτό ζητήσαμε τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Μάλιστα. Αυτά θα ακούσουμε σήμερα λοιπόν. Ευχαριστώ του τέσσερι εμπειρογνώμονε που είναι μαζί μα. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στο Γιώχαν Χόρν, που είναι εκπρόσωπος και επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης της Ingemetal στο Ingolstadt, και οι βουλευτές ε, διάβασαν το βιογραφικό σας γιατί υπήρχε στο φάκελο. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Funktioniert das αξιότιμη πρόεδρος, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, λέει ο κύριος Χόρν, να σας παρουσιάσω την άποψή μου σε αυτή τη δημόσια κρόαση με το θέμα ακριβώς ε, των διασυναριακών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου. Ε, υπάρχουν βεβαίως ε, πολυεθνικές, διασυνοριακές εταιρείες αν θέλετε, με διαφορετική υποδομή, με διαφορετική δομή και αρχιτεκτονική. Ε, αλλά υπάρχουν παραδείγματο χάρη εταιρείε που έχουν ίδια συστήματα παραγωγής και ίδιες εργασιακές ε, σχέσεις, ίδια πλαίσια. Χρησιμοποιούνται τα ίδια πρότυπα, οι ίδιες δομές για εσωτερική και εξωτερική ευελιξία και ε, παρόμοιοι μηχανισμοί ε, εφαρμόζονται διασυνοριακά στην Ευρώπη. Όλη η κουλτούρα των επιχειρήσεων που έχει διασυνοριακές ε, συναλλαγές υιοθετείται ακριβώς στις χώρες και στις τοποθεσίες όπου ενεργοποιείται αυτή η επιχείρηση δεδομένου ότι ακόμα και οι επικεφαλής managers προέρχονται από την έδρα, από τη μητρική εταιρεία. Αυτές ε, λοιπόν οι εταιρίες εταιρείες και η λειτουργία τους έχουν επιπτώσεις ε, ε, στις συνθήκες των εργαζομένων στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικοί κανόνες και ρυθμίσεις για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από την καθημερινή μου ζωή. Εγώ αντιπροσωπεύω από την ε, συνδικαλιστική μου ένωση 45.000 εργαζόμενους μετάλλου. Ε, είναι η εταιρεία Audi ΑΕ. έχουμε 28.000, η IG Metal, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση μετάλλου στη Γερμανία, έχει 28.000 εργαζόμενους από την Audi ΑΕ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας και θέλουμε να, να αναπτύξουμε περαιτέρω τις συλλογικέ μας διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμεθα στην Ουγγαρία. Εκεί φτιάχνουν ε, μηχανές αυτοκινήτων. Οι συνδικαλιστές συμφωνήσαν για λειτουργία αυτή διότι δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες απασχόλησης στην ε, Ουγγαρία και αυτή τη στιγμή ε, γίνεται όλη αυτή η μεταφορά του προγράμματος εργασίας της Σάουντι στην Ουγγαρία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή επεξεργαζόμαστε όλη αυτή τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας, παραγωγής. Και θέλουμε να εφαρμοστούν ήδη συνθήκες ε, διαχείρισης, management, εργασίας και λειτουργίας όπως στη Γερμανία, στη μητρική εταιρεία η επιχείρηση, η εταιρεία στην Ουγγαρία θα πρέπει να λειτουργεί όπως όλες οι άλλες εταιρείες στην Ευρώπη και να συμβάλλει ε, έτσι ώστε να γίνονται όλες ε, οι προσφορές για, για τον τρόπο εργασίας, ε, όλες οι, υποβάλλονται όλα τα προγράμματα, όλα τα project τα οποία θα εγκρίνονται από τη Μητρική στη Γερμανία. Και επίσης στο Βέλγιο υπάρχει άλλη μια εγκατάσταση παραγωγής της Audi ΑΕ. Η εταιρεία προσπαθεί να καθορίσει πρότυπα standards ε, για να εκμεταλλευτεί τις καλύτερες παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό προαπαιτεί βεβαίως ένα σταθερό ε, πλαίσιο ε, ε, εργασίας και παραγωγής και λειτουργίας. Αυτό όμως γίνεται σε κράτη τα οποία έχουν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Άρα λοιπόν οι μεγάλες διαφορές δεν είναι στην παραγωγή, είναι στις συνθήκες εργασίας, είναι στο εργασιακό πλαίσιο. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις μεγάλες εταιρείες αλλά και στους προμηθευτές. 20% Εμεί ε, εμείς έχουμε μια συμμετοχή 20% στην παραγωγή των ε, ε, προμηθευτών και 80% της προστιθέμενης αξίας προέρχεται από εκεί. Είτε είναι η Bosch, είτε είναι η Siemens, έχουμε συμβάσεις υπεργολαβίες και προμηθειών. Επίσης έχουμε και εταιρείε οι οποίες μέσα στα πλαίσια των εργαστικών συμβάσεων παρέχουν λογιστικές και προσωρινές εργασίες και καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι σε, με ίδιες συνθήκες δεν μπορούμε διασυνοριακά να εφαρμόσουμε ακριβώς τα ίδια πρότυπα, τα ίδια στάνταρτ σε διαφορετικές χώρες. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος εις βάρος των εργαζομένων εκμεταλλευόμενοι τις, περισσότερο, τις πιο αρνητικές συνθήκες εργασίας ή τα, χαμηλότερα στάνταρτ οι επιχειρήσεις αυτές να αντλούν ωφέλη εις βάρος των εργαζομένων. Παραδείγματο χάρη, εξέτοντους σε κινδύνους ε, που αυτά δεν γίνονται στη μητρική εταιρεία, στην χώρα της έδρας, ε, μειώνοντας ε, τις, τις απολαβές και άλλα τινά. Εμείς ε, προτείναμε λύσεις σε αυτό, κάναμε μία μελέτη και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο στάθμισης. Ε, δεν θέλουμε οι εργαζόμενοι για να εξασφαλίσουν την εργασία τους, να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις τους και να δεχθούν χαμηλότερες και χειρότερες συνθήκες εργασίας και ε, ε, με την εξασφάλιση υποτίθεται της δουλειά τους. Γίνεται λοιπόν ένας φαύλος κύκλος μεταξύ προσφοράς αλλά και χαμηλότερων, ε, παροχής χαμηλότερων δικαιωμάτων. Θέλουμε να Θέλω να αναφερθώ τώρα στις ε, υποχρεωτικές ε, διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους, τις οποίες ρυθμίζει η οδηγία ε, των εργασιακών συμβουλίων. Όλες αυτές οι δυνατότητες δίνονται στους εργαζόμενους και για την πράσπιση των συμφερόντων τους λειτουργούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτές προάγουν τα δημοκρατικά συμφέροντα των εργαζομένων, έστω και υπό διαφορετικές συνθήκες και βεβαίως διασυνοριακά. Ε, αν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις οργανώσεις, στα συνδικάτα αυτά, μπορούν να λαμβάνουν μέρος και στις διαπραγματεύσεις μέσω των εκπροσώπων τους, στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Θέλουμε εμείς να εδραιώσουμε μία ενιαία, ένα ενιαίο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων με διαφορετικές, ε, σε χώρες με διαφορετικές συνθήκες. Μία κουλτούρα δηλαδή, θέλουμε να είναι ομοιόμορφη και ενιαία η κουλτούρα αυτή, η οποία να είναι και επιχειρησιακή αλλά και ευρωπαϊκή. Και επειδή θέλουμε να είναι ευρωπαϊκή πρέπει οπωσδήποτε να είναι και δημοκρατική. Πώς μπορούμε λοιπόν να καλεί συνθήκες διαφορετικά πρότυπα σε ένα πλαίσιο. Αυτά θα πρέπει να, υπά... να τα έχουμε υπόψη μας κάθε φορά που γίνονται συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θεμητή διαπραγμάτευση λοιπόν και δίκαιη. Αυτή να πετούμε. Όχι για να οξύνουμε τον ανταγωνισμό, αλλά για να επιτύχουμε την καλύτερη ε, παραγωγή, τα καλύτερα προϊόντα, το καλύτερο αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές αν βελτιωθούν ε, τα προϊόντα, αν υπάρχει το ποιοτικό στοιχείο, αν υπάρχει καλή παραγωγή, σαφώς αυτό ε, ενεργεί προς όφελος των εργαζομένων. Ο λόγος τώρα στον κύριο Ρικάρντο Ροντρίγκε, που είναι Ισπανός, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης Ένωσης των ε, Εργαζομένων. Κύριε Ροντρίγκε, για 7 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου σύστησαν να μιλάω, να μιλήσω λίγο, δυνατά και καθαρά. Το λίγο σίγουρο, διότι δεν μου δίνεται και πολύ χρόνο. Αυτή η ακρόαση είναι για να δώσουμε την άποψή μας στον εισηγητή. Οπότε θα είμαι τηλεγραφικός. Τέσσερα σημεία πρέπει να θίξουμε. Πρώτον, ο τίτλος της έκθεσης ε, δείχνει ότι έχει σχέση στην πραγματικότητα με την ερώτηση αν θα πρέπει να υφίσταται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων. Πιστεύω ότι από την αρχή τη δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την αρχή της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Εκτιμένου σε εργασιακά θέματα έχουμε κάνει πολύ μεγάλο, πολύ μακρύ δρόμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορους φορείς που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αντιπροσωπευτικοί και που δρούν σε διάφορα επίπεδα. Και στον ε, κλαδικό τομέα, ε, όσο και κλαδικά. Υπάρχουν επίσης διάφορες διαδικασίες διαλόγου που καταλήγει σε διαφόρων ειδών συμφωνίες, κλαδικές, τομεακές, ευρωπαϊκές κλπ. Σύμβολα υπάρχουν πολλές διαδικασίες, πολλές συμφωνίες και πολλοί φορείς. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι ένα σύστημα. Και τι λείπει για να έχουμε αυτό το σύστημα. Δύο πράγματα. Πρώτον, η δυνατότητα αυτές οι συμφωνίες να είναι υποχρεωτικές, δεσμευτικές και εφαρμόσιμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλων των ειδών της εργασιακές σχέσεις, που είναι πολλές, και δεύτερον, μια ισοδυναμία ε, και ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό χώρο επίλυσης διασυνοριακών διαφορών εργασιακών σχέσεων ένας ε, χώρος ο οποίος δεν θα είναι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι ένας ε, χώρος ο οποίος θα, έχει ως στόχο την επίλυση, προληπτική ε, επίλυση εργασιακών διαφορών, μη δικαστικών διαφορών. Ε, δεύτερον, κάτι το οποίο τίνουμε να αμελούμε. Τι σημαίνει διαμεθοριακός, διασυνοριακός. Μιλούμε για διασυνοριακό κοινωνικό διάλογο, για, ε, για συλλογικές διαπραγματεύσεις διασυνοριακές κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το διασυνοριακό. Γιατί το διασυνοριακό θα μπορούσε να είναι υπερεθνικό, θα μπορούσε να είναι διεθνές. Θα μπορούσε να σημαίνει cross-border, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την αγγλική λέξη, transfrontalier γαλλικά, για μένα το διασυνοριακό σε ένα ενδεχόμενο σύστημα συλλογική διαπραγμάτευση ή επίλυσης, εξοδικαστική επίλυση διαφορών ε, έχει κάποια συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες ελάχιστε απαιτήσει και χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι θα πρέπει να επηρεάζει πάνω, άνω του ενό κράτη-μέλη. Τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη, δηλαδή, με λίγα λόγια. Δεύτερον, δεύτερη απέτηση, δεύτερο όρο, να εμπλέκεται μια επιχείρηση σε κοινοτικό επίπεδο, κοινοτικής κλίμακος ή να εμπλέκονται δύο περισσότερες επιχειρήσεις, έστω και σε εθνικό επίπεδο, που όμως αποτελούν τμήμα ενός συγκεκριμένου οικονομικού κλάδου ή τομέα. Ε, αυτός ο ορισμός έχει σχέση με τους κοινωνικούς εταίρους ε, που εμπλέκονται. Τώρα, αυτές είναι ελάχιστες απαιτήσει. Από εκεί και πέρα μπορούν να προσθεθούν και άλλα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, συλλογικές, ε, διασυνορικές συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν, που είναι περιφερειακής φύσεως. Εργασιακές σχέσεις που, ε, ρυθμίζουν εργασιακές σχέσεις σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Τρίτον, γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό ή διασυνοριακό, αν θέλετε, εργασιακό, πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή σε αυτή την περίπτωση διασυνοριακών συλλογικών συμβάσεων. Πρώτον, διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κοινωνικός κλαδικός διάλογος, η διασυνοριακο αν θελετε εργασιακο πλαισιο εργασιακων σχεσεων η σε αυτη την περιπτωση διασυνοριακων συλλογικων συμβασεων πρωτον διοτι υπαρχουν ενδειξει οτι ο κοινωνικος κλαδικος διαλογος η αποτελεσματικοτητα του σε εθνικό επίπεδο είναι αμφισβητήσιμη. Μιλώ για τον κλαδικό κοινωνικό διάλογο και τις συμφωνίες οι οποίες δεσμεύουν τους υπογράφοντες. Ε, αυτές οι συμφωνίες ε, πραγματικά υπολείπονται του επιθυμητού. Επίσης, είναι απαραίτητο να συνεισφέρουμε στο να ε, βελτιώσουμε, να συμπληρώσουμε την εσωτερική αγορά. Ε, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα θα επέτρεπε να συμπληρωθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. Για παράδειγμα, θα, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα θα είχε ωφέλη για την πρόληψη ε, εργασιακών διαφορών, διασυνοριακών εργασιακών διαφορών, κάτι που θα μας οδηγούσε σε εξοικονόμηση χρόνου, πόρων, φόρτου Καθώς επίσης, όπως αναφέρει και ο εισηγητής, θα μας επέτρεπε ένα τέτοιο σύστημα να αντιμετωπίσουμε καινούργια φαινόμενα τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη πλειοψηφία. Πλην όμως είναι σημαντικά, ε, μιλούμε για συμφωνίες μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων που ε, μπορεί να είναι ενδεικτικές προς το παρόν, πλην όμως ε, όλο και περισσότερο ρυθμίζουν ε, εργασιακές σχέσεις, συνθήκες εργασίας που ε, αρχίζουν να μοιάζουν με πραγματική διασυνορική ε, διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων. Τέταρτο σημείο. Ε, Πώ θα μπορούσαν να λάβουν χώρα αυτέ οι συλλογικέ διαπραγματεύσει σε διασυνοριακό επίπεδο. Θα, εστιαστώ, θα εστιάσω σε επίπεδο επιχείρηση, διότι για το κλαδικό επίπεδο νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου έχουν να πούν περισσότερα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, Υπάρχουν τέσσερα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε ε, διασυνοριακή συλλογική διαπραγμάτευση. Πρώτον, ένα από τα βασικά εμπόδια ήταν πάντοτε να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί που διαπραγματεύονται, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπογράφουν είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει εμείς που ε, μελετούμε σε βάθος όλες τις, ε, σχεδόν όλες τις δυνατότητες και τα σενάρια ε, τα οποία θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε διάφορους φορείς, επιτρο, ευρω, επιτροπές επιχείρησης, Ευρωπαϊκών, Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχείρησης, ομοσπονδίες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργοδοτών και εργαζομένων και βέβαια συνομοσπονδίες που σε εθνικό επίπεδο που θα μπορούσαν να υπογράψουν ε, τις ευρωπαϊκές συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις ε, συμφωνίες προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές συλλογικές διαπραγματεύσεις και μάλιστα θα μπορούσαν να διευκολύνουν και την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο. Τελειώνοντας, θα έλεγα ότι έχουμε δύο ακόμα πτυχές. Πρώτον, την σύνδεση με το, ε, το κλαδικό επίπεδο. Αυτά ήταν που ήθελα να πω στον εισηγητή. Κατά βάση θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια να συμπληρωθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων. Αυτή η δυνατότητα θα έπρεπε να αρχίσει να συζητείται ήδη ε, οι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Οποιαδήποτε λύση ε, επιλεγεί πιστεύω θα πρέπει να όσο πιο ευρωπαϊκή γίνεται γιατί θα έχει λιγότερα προβλήματα στην εφαρμογή της. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ε, και θα ήθελα το τελικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί ε, το, το αν θα είναι δηλαδή νομικής ή μη νομικής φύσεως θα έπρεπε να συζητηθεί τελευταίο. Και όπως είπε και ο εισηγητής, υπάρχει κι άλλο ένα θέμα για άλλη ακρόαση. Ποιο είναι το, ποιες είναι οι, ποιος είναι ο αντίκτυπος συγκεκριμένων αποφάσεων του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την άσκηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στον τρίτο προσκεκλημένο, ο κύριος λούτ Μιούλ, Διευθυντής Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Ευθύνης, Κοινωνικού Ευρωπαϊκού ή διεθνούς διαλόγου στην Γερμανική Οργάνωση Εργοδοτών Χημικών Βιομηχανιών. Έχετε 7 λεπτά, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, κύριε Νούγλα. Αξιότιμοι πρόεδρος, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιάσω τη θέση μου σε αυτή την ακρόση και είναι μια εξαιρετική ιδέα που ως εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων μπορούμε να συζητήσουμε τις ενδεχομένως αντίθετες απόψεις μας. Ε, δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Πρώτον, είμαι εκπρόσωπος ε, της, της Γερμανικής Ομοσπονδίας εργαζομένων στη χημική βιομηχανία, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι υψηλών προδιαγραφών και δεξιοτήτων. Και αμείβονται σχετικά με τους άλλους εργαζόμενους πολύ καλά. Βεβαίως η εργασία τους εμπεριέχει και ορισμένους κινδύνους. Ας πούμε τα βαρέα και ενθυγιεινά, όπως λέμε. Είμαστε λοιπόν πεπισμένη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της εταιρική διαδικασίας και όλο αυτό το πλαίσιο έχει δώσει εξαιρετικά καλά αποτελέσματα στη Γερμανία έχουν ε, συμπεριληφθεί, έχουν συγγνώμη, συμπεριφερθεί και οι δύο πλευρές πάρα πολύ καλά, με πολύ καλή θέληση και βούληση συνεργασία και τις τελευταίες δεκαετίες στη Γερμανία έχουμε εδραιώσει έναν επιτυχημένο διάλογο με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μακάρι να μπορούσε αυτό το πλαίσιο να εφαρμοστεί και σε διεθνές επίπεδο. Όταν βεβαίω γίνονται διασυνοριακέ ε, συλλογικέ διαπραγματεύσει, ένα διασυνοριακό κοινωνικό διάλογο, είναι πολύ σημαντικό να, ακολουθήσουμε, να παρακολουθούμε το πλαίσιο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών Ευρωπαϊκών Εργασιακών Συμβουλίων. Αυτό έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν βεβαίως ε, ε, ένα κοινό πλαίσιο αντιλήψεως, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές αντιλήψεις. Ε, όλα αυτά ακούγονται ωραία, αλλά ε, δεν θέλω να ωρεοποιήσω υπερβολικά και να πλουστεύσω το θέμα, διότι είναι περίπλοκο. Παρόλα τα ωραία και θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές προκλήσεις. Και αυτές οι προκλήσεις οφείλονται κυρίως στα διαφορετικά συστήματα κοινωνικών σχέσεων που υπάρχουν ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι γεγονός. Ε, δεν είναι η θέση μας να το κρίνουμε. Όμως αυτοί, αυτές οι διαφορές ε, είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν δύσκολες καταστάσεις στην Ευρώπη. Ε, διαφορές, ε, η ευθύνη και τα λάθη δεν ε, μπορούμε να τα φορτώσουμε ούτε στους εργοδότες, ούτε στους εργαζόμενους, ούτε στις κοινωνικές συνθήκες. Εδώ έχουμε στην Ευρώπη διαφορετικές ιστορικές εξελίξεις που είτε μας αρέσει είτε όχι έχουν οδηγήσει σε μια διαφορετική κοινωνική κατάσταση, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικό εργασιακό δίκαιο κλπ. Δεν μπορούμε λοιπόν να απαιτούμε ένα απόλυτα εναρμονισμένο σύστημα σύστημα να λαμβάνουμε υπόψη τις, διαφορο... τις αυτές. Τώρα, αν θέλετε να, να επιδιώξετε μια τέτοια εναρμόνιση, θα πρέπει καταρχάς να εδραιώσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη, δηλαδή πώς φανταζόμαστε όλοι ομοιόμορφα και ενιαία ένα πανευρωπαϊκό σύστημα, ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα, είμαι οπαδός ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου και έχω συμμετάσχει και ε, δραστήρια τα τελευταία δέκα χρόνια και έχω μια σαφή εικόνα στα, σε πολλά κράτη-μέλη. Αλλά δεν έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει αυτή η βούληση της πλήρης, πλήρους ομοιομορφίας και της πλήρους εναρμόνισης των εργασιακών σχέσεων και των συστημάτων. Πάντοτε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, πάντοτε οι, κοινωνι... οι σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων θα, είναι... θα έχουν το στοιχείο της δυσκολίας, θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει και το στοιχείο της ευελιξίας, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως έχει στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το συμπέρασμά μου είναι η εξής, ότι προς το παρόν σε εθνικό επίπεδο το εθνικό επίπεδο είναι το καθοριστικό για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Ε, λειτουργεί μέσα σε ένα ορθολογικό πλαίσιο. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει. Ε, σε αυτό το επίπεδο το εθνικό καθορίζονται οι συνθήκες εργασίας, το ωράριο, η μισθοί, οι απολαβές κλπ και δεν είναι δυνατόν να εναρμονίσουμε όλο το σύστημα στα 27 κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι τα Ευρωπαϊκά Εργασιακά Συμβούλια λειτουργούν θαυμάσια, είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για να βοηθήσουν τις λογικές διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τώρα αυτά που είπε ο εισηγητής προς συζήτηση, θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου οι εργαζόμενοι έτσι κι μέσα στα Ευρωπαϊκά Εργασιακά Συμβούλια λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, λειτουργούν ικανοποιητικά, λειτουργούν επαρκώς και δεν είναι δυνατό να κατηγορήσετε από την πλευρά δηλαδή, των εργαζομένων ότι δεν ενημερώνεται και δεν υπάρχει πληροφόρηση. Ε, άρα πολλές εταιρείε έχουν, αναβι... Ε, έχουν προάγει... προαγάγει αυτά τα εργασιακά συμβούλια σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο έτσι ώστε να λειτουργούν πραγματικά ε, πολύ, πολύ ικανοποιητικά και πολύ καλά. Ε, δεν είναι δυνατόν να, να καταργήσουμε ή να μειώσουμε τα, τα ε, τα ελάχιστα πρότυπα επί καθημερινής βάσης, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατηγορήσουμε ε, τους, ε, την, την πλευρά της εργοδοσίας για μία πληροφόρηση για την έλλειψη ενημέρωσης, δεδομένου ότι μέσω των εργασιακών συμβουλίων έχουμε επιτύχει ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πιστεύω ότι η λύση είναι περισσότερες κανονιστικές ρυθμίσεις, περισσότεροι κανονισμοί, περισσότερο βάρος της κανονιστικής πλευράς. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαυμάσια τα εργαλεία που έχουμε. Ε, πρέπει να πείσουμε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης εκεί όπου δεν συμμετέχουν. Τώρα, για τις ε, διασυνοριακές συμφωνίες, διασυνοριακές ε, συλλογικέ ε, συλλογικές συμβάσεις, αυτές δεν ορίζονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ορίζονται από τους συμμετέχοντες, από τα δύο μέρη που συμμετέχουν. Αυτές οι συμφωνίες δεν είναι μαζικό φαινόμενο. Τουλάχιστον στη Γερμανία κάτω από το 1% των επιχειρήσεων υποχρεούται να ε, υπογράψει διασυνοριακές συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις. Αυτές λοιπόν οι συμφωνίες, οι διασυνοριακές αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό όλων των ε, πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται και πάλι εδώ για τον, την υποχρέωση σεβασμού πολύ διαφορετικών κανονισμών ε, οι οποίες διασυνοριακές συμφωνίες υπογράφονται από τις εταιρείες χωρίς να έχουν καμία επίπτωση ε, στο κρατικό επίπεδο, ούτε το κρατικό επίπεδο να έχει επίπτωση σε αυτές. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία έντολη να αλλάξει η κατάσταση αυτή και να παρέμβει είτε το εθνικό είτε το ευρικό επίπεδο. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα στις ε, διασυνορικές ε, συλλογικές πραγματεύσεις και τις κοινωνικές σχέσεις. Ο στόχος μας είναι να συζητήσουμε κάθε προτινόμενη ιδέα με επικοδομητικό πνεύμα και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει διόλου ανάγκη περαιτέρω ευρωπαϊκής ρύθμισης ε, ή η παρέμβαση στις διασυνοριακές συμφωνίες που κάνουν οι εταιρείε. Αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε στο εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο εργασιακού συμβουλίου είναι επαρκέστατο και λειτουργεί θαυμάσια. Περαιτέρω παρεμβάσεις δεν χρειάζονται. Θα δούμε τι θα δώσει η συζήτηση που θα λάβει η χώρα μετά, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον τελευταίο προσκεκλημένο, που τον ευχαριστώ που ήρθε, που είναι ο Στέφαν Κολινιό, που είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας στη Σχολή Σπουδών Σαντάνα, στην Πίζα, και ήταν επίσης καθηγητής στο Χάρβαρντ και στο London School of Economics. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, δύο πράγματα. Σε 7 λεπτά μπορείτε να πείτε πολλά, αλλά δεν μπορείτε να αποδείξετε τίποτα. Ε, γι' αυτό έγραψα ένα κείμενο αρκετά μακροσκελές, το έχετε μπροστά σας και σας δίνει και κάποια στοιχεία που συμπληρώνουν αυτά που θα πω προφορικά. Ε, δεν εκπροσωπώ κανένα, κανένα λόμπι, καμία οργάνωση, είμαι ακαδημαϊκός και επομένως ως ακαδημαϊκός θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο αυτή τη συζήτηση και αντί να εξετάσουμε ε, τους συντελεστές ε, της διαπραγμάτευσης για τα μισθολογικά, να δούμε το αποτέλεσμα. Και κυρίως να αναλύσουμε τις επιπτώσεις ε, της διαδικασίας για την α, μακροοικονομικές ανισορροπίες και τη διαδικασία εξυγίανσης που έχουμε που βλέπουμε και ζούμε στην ευρωπαϊκή κρίση και τη σημαντική διαδικασία προσαρμογής που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Οι διαπραγματεύσεις για τα μισθολογικά είναι βασική μεταβλητή, γιατί καθορίζει τις ε, την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και τα πλεονεκτήματα περιφερειακά και ένας τρόπος να προσελκύσουμε επενδύσεις. Η ανταγωνιστικότητα, μάλιστα, είναι οι προποθέσει υπό τις οποίες μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Είναι πολύ γνωστό ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας ε, τροποποιήθηκε από το 2008 μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το είπε πολλές φορές και πολλοί άλλοι ερευνητές ε, και υπεύθυνοι το είπαν επίσης. Από το 2008 επίσης ε, είδαμε ότι τουλάχιστον στις χώρες που πλήρονται πολύ από την κρίση στην Νότια Ευρώπη αυτή η τάση έχει αντιστραφεί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αν δούμε τους ε, λόγους πίσω από αυτή την προσαρμογή θα δείτε ότι έχουμε, όταν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα μισθολογικά σημαίνει ότι οι αλλαγές, οι ονομαστικές αλλαγές ε, στους μισθούς ήταν πιο σημαντικές από την παραγωγικότητα. Κατά την κρίση αυτοί οι ονομαστικές οι ονομαστικοί μισθοί ας πούμε στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα έπεσαν αλλά πολύ ενδιαφέρον άρχισαν να αυξάνονται πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη στη Γερμανία. Αυτό που προκάλεσε αυτή την αλλαγή είναι το εξής. Ε, Έχουμε συντονισμένες διαπραγματεύσεις για τα μισθολογικά. Όχι. Ε, πανερχόμαστε στην ε, ε καμπύλη Φίλιπς. Μέχρι το 2008 δηλαδή η αύξηση των μισθών δεν ε, ανταποκρινόταν ή δεν αντικατόπτριζαν τις ε, αλλαγές στην απασχόληση και στην ανεργία και εστιάζονταν κυρίως στην παραγωγικότητα και σε εξελίξη παραγωγικότητας. Όμως από το 2008 ε, βλέπουμε ότι η απασχόληση και κυρίως ε, η μείωση της απασχόλησης, δηλαδή η ανεργία, ε, ήταν πολύ σημαντική για τον καθορισμό των μισθών εκ νέου. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε ε, ουσιαστικά ένα οικονομικό μηχανισμό εντελώς προσαρμοσμένο στην αγορά, αλλά δεν έχουμε κανένα συντονισμό και καμία πολιτική ή κανένα εργαλείο πολιτική εν για την προσαρμογή. Παρενέργεια αυτού που είναι ενδιαφέρουσα και διαφορετική από αυτά που, αυτό που θα περιμέναμε είναι ότι η κερδοφορία στην Ευρωζώνη συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής με την εξαίρεση της Ιρλανδίας, Ισπανίας, ε, ε, Πορτογαλίας και Ελλάδας. Αυτά τα περιθώρια κερδοφορίας, όπως προκύπτει από τις ε, διαδικασίες διαπραγματεύσεων για τα μισθολογικά σημαίνει ότι οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν λιγότερο από την παραγωγικότητα. Αν κοιτάξετε την ανταγωνιστικότητα με ευρύτερου όρου, είναι σημαντικό να εξετάσουμε και την, τα κέρδη των κεφαλαίων. Πέρα από την παραγωγικότητα της εργασίας και τον καθορισμό των μισθών, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παραγωγικότητα των κεφαλαίων. Εδώ βρίσκουμε ότι τα κέρδη των κεφαλαίων σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο έχουν βελτιωθεί στην Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, έχουν επιδεινωθεί στην Ολλανδία, Φιλανδία και στη Γαλλία, έχουν παραμείνει περίπου σταθερά με μικρές διακυμάνσεις στη Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον καθορισμό μισθών σε εθνικό επίπεδο που μίλησαν για αυτά οι προηγούμενοι ομιλητές και είπαν ότι είναι σημαντικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης για τα μισθολογικά. Αλλά σημαντικό είναι να δούμε και τις ε, κλαδικές προσαρμογές ε, ανάμεσα στους ε, τομείς του εμπορίου και τους τομείς που δεν είναι του εμπορίου. Ο Κάνφορς και Τρίφελ πριν από λίγα χρόνια είπαν ότι οι διαπραγματεύσεις για τα μισθολογικά σε, στις δύο ακραίες περιπτώσεις πολύ συγκεντρωτικό σύστημα ή αποκεντρωμένο σύστημα είναι βέλτιστο ε, μακροοικονομικά, αλλά ε, είναι προβληματικό ε, στο εσωτερικό. Δηλαδή με τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που, έχει, που, που είναι λίγο υβριδικό. Το συμπέρασμα είναι ότι οι στραβλώσεις που είχαμε πριν από το 2008 εξακολουθούν να ισχύουν ε, και να επαυξάνονται. Ε, υπάρχουν τρία κανάλια προσαρμογής που έχουμε σε αυτό το πλαίσιο για το, ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Το ένα είναι η μισθή, το άλλο είναι τα κέρδη και το άλλο είναι οι τιμές. Και αυτές οι προσαρμογές, αν λάβουν χώρα τομεακά, κλαδικά, αυτό σημαίνει ότι αν κοιτάξουμε και τους τομείς που δεν έχουν σχέση με το εμπόριο και την προσαρμογή των μισθών, ε, αυτή η προσαρμογή των μισθών ε, είναι το κανάλι μέσα από το οποίο γίνεται η, προσαρμογή. η προσαρμογή. Οι τομεί τη οικονομία που δεν συνδέονται με το ενιαίο νόμισμα, που δεν συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, αισθάνονται ότι πλήττονται. Από την άλλη, οι τομεί που δεν έχουν σχέση με το εμπόριο, με μικρότερε αυξήσει στι την παραγωγικότητα, που όταν υπάρχει προσαρμογή μέσω των ε, κερδών, εκεί βλέπετε ότι οι εταιρείε, επειδή μειώνεται ε, το περιθώριο των κερδών, τους παραπονιούνται. Έτσι, είτε έχουμε ευρωσκεπτικισμό και ευρωσκεπτικιστικέ τάσει πολιτικά ή αλλιώς έχουμε ε, αριστερό ευρωσκεπτικισμό αν έχουμε συμπίεση των μισθών ή δεξιό σκεπτικισμό ανάλογα με το επίπεδο των μισθών. Και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση που η προσαρμογή είναι μέσω των τιμών, έχουμε ότι το, το αποτέλεσμα Σάμιουσον είναι αυτό που ισχύει στην Ευρωζώνη για την ε, Γαλλία και την Ιρλανδία, όπου οι μισθοί έχουν μειωθεί, ενώ στην Ιταλία και στην Ελλάδα περίπου και έχουν μειωθεί επίσης, ενώ παρέμειναν σταθεροί στην Ισπανία και κάτι που δεν περιμέναμε ε, για μια αγγλοσαξονική οικονομία στι ε, ΗΠΑ. Στην Ιταλία αυξήθηκαν τα κέρδη για του τομεί που δεν έχουν σχέση με το εμπόριο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στην Ισπανία παρέμειναν σταθεροί, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι ΗΠΑ έπεσαν ε, κατά τη διάρκεια τη κρίση. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει μια ανάγκη να συντονίσουμε πιο έντονα τους διάφορους τομείς και να δούμε ποιος παίζει τον ηγετικό ρόλο Ποιο καθορίζει ε, τους μισθούς, κάνει τι διαπραγματεύσει, ε, πρέπει να δείξουμε τι γίνεται με του τομεί που εξαρτώνται από το εμπόριο και αυτού που δεν εξαρτώνται. Η Βόρεια Ευρώπη πριν από την κρίση, όπω λέει το έγγραφό μου, εστίασε κυρίω σε χαμηλότερε αυξήσει των μισθών στου βιομηχανικού τομεί, ενώ ο Νότο ήθελε ψηλότερες, ε, είχε αυξήσεις ε, των μισθών στις ε, υπηρεσίε. Τώρα, για τα καθεστώτα διαπραγμάτευση για τα μισθολογικά. Ποιε είναι οι επιπτώσει, Έχουμε ε, διαπραγματεύσει σε επίπεδο πολυεθνικών. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Που δεν αρκούν όμω πια, ούτω ώστε να έχουμε συντονισμό των μισθό που να συνάδει με το χώρο τη Ευρωζώνη, του ενιαίου νομίσματο. Ε, Μία συνεκτική προσέγγιση για τον τομέα τη Ευρωζώνη σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την παραγωγικότητα της εργασίας, του κεφαλαίου και την ε, κατανομή ανάμεσα στο, στην εργασία και στο κεφάλαιο, καθώς και μεταξύ των περιφερειών, χωρών και τομέων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε το διακλαδικό στοιχείο, αλλά και το ενδοκλαδικό στοιχείο και, εκεί, και να συντονίσουμε και στα δύο επίπεδα τους μισθούς. Δεύτερον, μακροοικονομικός διάλογος, ο οποίος ε, ξεκίνησε το 1999. Αυτός απέτυχε, όπως είδαμε από τις ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν και ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι οι Υπουργοί Οικονομικών και, κοινωνικό, και οι κοινωνικοί εταίροι έκαναν τα δικά τους και αυτοί ασχολούνταν. Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς το εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δίνετε κι εσείς ε, μηνύματα προς αυτούς. Επίσης, ένας κανόνας για τους μισθούς δέχτηκε, έγινε δεκτός ε, γενικά. Ότι η ονομαστική αξία των μισθών θα πρέπει να συνάδει με την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Μπορεί να αρκεί στα μάτια της ΕΚΤ, αλλά δεν αρκεί για να σταματήσουμε τις ανισορροπίες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 12 λεπτά διερμηνίας ακόμα. Ε, τρεις ομιλητές, σύντονοι συγητή τέσσερις ε, πρέπει να δώσουμε χρόνο και στους καλεσμένους μας να απαντήσουν, οπότε περιοριστείτε σε δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Μωρέν Σαρτιέ και μετά ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Σε αυτή την περίοδο κρίσης που διερχόμαστε αντιλαμβανόμαστε ότι τρία ζητήματα ε, σηματοδοτούν τον κοινωνικό διάλογο και το χαρακτηρίζουν. Πρώτον, ανάγκη ε, οικοδόμησης μιας κοινωνικής συνοχής μεταξύ των 27, ε, οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης, πολύ περίπλοκο, δεδομένων των διάφορων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεν θα μπω σε αυτό το ζήτημα. Δεύτερο χαρακτηριστικό ε, που μας ανησυχεί είναι η, εξέλιξη της απασχόλησης, κοινωνικός διάλογος, αλλά οπωσδήποτε στόχος μας είναι η αύξηση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης και η προσαρμογή τους ε, στα καινούργια δεδομένα και καινούργιες απαιτήσεις και εδώ χρειαζόμαστε κοινωνικό διάλογο και κινητοποίηση όλων και τρίτο σημείο πολύ σημαντικό το να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Κοινωνικός διάλογος λοιπόν γίνεται και για να επιτευχθούν και οι τρεις αυτοί στόχοι. Κοινωνική συνοχή, αύξηση της απασχόλησης και αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ε, Ευχαριστώ, Όλε Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους καλεσμένους μας ε, για τις, ε, τη συμβολή τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε την άποψη των εργαζομένων. Βεβαίως θέλουμε κοινωνικός ε, διάλογο να διέπεται από κανόνες και να μην μπορούν αλλά και οι εργοδότες να μπορούν ε, να ε, χειρίζονται τα θέματα που θέλουν ε, μέσα στα πλαίσια του θεμητού ανταγωνισμού. Όλοι εάν βεβαίως όλοι οι πολίτες μας έχουν εργασίες μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και με τις οικογένειές τους ε, και να επιλέξουν και μάλιστα με τη χώρα, τη χώρα στην οποία θέλουν να ζήσουν που έχει φθηνότερο κόστος διαβίωσης. Γι' αυτό η αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική και οι συνθήκες ε, βάσει των οποίων λειτουργούν. Ε, βλέπετε ότι εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου μία μεγάλη εταιρεία, τεράστια εταιρεία μεταφέρει όλη την παραγωγική της υποδομή σε μία άλλη χώρα και όλα τα συστήματα παραγωγής τα μεταφέρει ως έχουν από την μητρική χώρα στην καινούργια χώρα εγκατάστασης. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ε, μία, τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και μισθοδοσίας των υπαλλήλων να, να παίρνουν τον, έναν μισθό που τους επιτρέπει να ζουν καλά, ε, να αμείβονται δίκαια. Ε, καταλαβαίνω βεβαίω ότι πολλές χώρες προσπαθούν να προσφέρουν κίνητρα για να προσελκύσουν ακριβώς αυτή τη μεταφορά ε, λειτουργία εταιριών. Και η, ακριβώ η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η έκθεση Χέντελ είναι ιδιαίτερα σημαντική μια στιγμή που μιλούμε για εμβάθυνση της ε, ΟΝΕ και συζητούμε για την προσθήκη ενός ε, κοινωνικού πυλώνα στην ΟΝΕ. Αυτό είναι υποσυζήτηση, αλλά προφανώς εκκρεμεί. Καταλαβαίνω λοιπόν την ανάγκη σεβασμού των ε, εθνικών πρακτικών και των εθνικών παραδόσεων. Όμως, αν δεν μετακινηθούμε κιόλας, η κοινωνική εταίροι και οι εργαζόμενοι τελικά θα πληρώσουν την ύφη. Ο Στεφάν Κολινιό το εξήγησε. Τιμές, μισθή, κέρδη μας επιβάλλουν να λάβουμε υπόψη την, τον οικονομικό μας περίγυρο, την οικονομική συγκυρία. Ε, ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, έχω εκπλαγεί σε δύο περιπτώσεις που εξετάσαμε ε, πρακτικά τις ε, συνθήκες ε, του διασυνορακού διαλόγου για, όταν χρησιμοποίησαμε το Ταμείο Βοήθειας για την Όκια και την ΤΕΛ, το Ταμείο ε, στην Παγκοσμιοποίηση. Η ΤΕΛ παρήγαγε ε, υπολογιστέ στην Ιρλανδία και με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κρατικές ενισχύσεις μετακινήθηκε στην Πολωνία για, ε, τους, για να παράγει εκεί ε, ε υπολογιστές. Ε, η, η είχε 2.000 εργαζόμενους χωρίς συνδικαλισμό. Ε, η Dell, συγγνώμη, είχε 2.000 εργαζόμενους χωρίς συνδικαλισμό καθόλου. η Νόκια έκλεισε στη Γερμανία για να ανοίξει στην Ρουμανία και μετά έκλεισε στη Ρουμανία για να πάει στην Κίνα πριν καν να κλείσει το εργοστάσιό της στη Ρουμανία. Και στην Στρογγυλή Τράπεζα για την Χαλιβουργία που ε, ε, οργάνωσε ο κύριος Ταγιάννη την περασμένη εβδομάδα, ε, ο Επίτροπος άνοιξε τη συζήτηση ζητώντας την, από την Αρσελόρ Μιτάλ να αναστείλει το κλείσιμο του εργοστασίου της μέχρι να υποβάλει προτάσεις ο ίδιος και η απάντηση της Μιτάλ ήταν η Κομισιόν πρέπει να μας βοηθήσει να, κατα, να ε, καταπολεμήσουμε ε, την ε, ε φοροδιαφυγή στην ε, Πολωνία γιατί αλλιώς θα χρειαστεί να κλείσουμε. Έχουμε δύο διαφορετικές λοιπόν προσεγγίσεις που μας ξεπερνούν. οπότε θα ρωτούσα τους φιλοξενούμενους μας ε, τι θα πιστεύατε για την δημιουργία ε, τη, ενός σώματος Ευρωπαίων Ευρωπαϊκών ελεκτών Εργασίας, από, που θα προέρχονται από διάφορες ε, ε, χώρες και διάφορες παραδόσεις και ποιοι είναι οι όροι μέσω οποίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος. ο μακροοικονομικός διάλογος ε, στο περιθώριο του Συμβουλίου Δεκεμβρίου δεν χρησιμεύτηκε σε πολλά πράγματα. Ζητώ, συγγνώμη που ξέπαρασα το, το χρόνο μου. Δίνω το λόγο στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες για το χρόνο που μας έδωσαν για αυτή τη συζήτηση. Η περιπλοκότητα τονίστηκε και πάλι. Αλλά λάβαμε ισχυρές ενδείξεις για το τι μπορούμε να διευθετήσουμε στο μέλλον. Και δει εγώ συζητητής. Εδώ δεν πρόκειται να εναρμονίσουμε, να δημιουργήσουμε ομοιόμορφες ε, ρυθμίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι οράματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα χειριστεί το Κοινοβούλιο. Όμως υπάρχουν και συνθήκες τις οποίες δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Θέλουμε να εδραιώσουμε ένα εργασιακό πλαίσιο το οποίο να τηρεί και να σέβεται τον ευρωπαϊκό διάλογο, ε, το ευρωπαϊκό κανονιστικό ε, πλαίσιο και να αποφύγει τριβές και παραβιάσεις. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να συνεργαστούμε την Κομισιόν και μετά από τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων ε, μας βοηθούν όλες αυτές οι απόψεις και θα ε, στείλω και την έκθεση η οποία υιοθετήθηκε πέρσι ε, για ένα παρόμοιο θέμα στη Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων. Ε, πιστεύω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με περισσότερα στοιχεία, με περισσότερα επιχειρήματα και ελπίζουμε να τύχουμε μια ευρεία υποστήριξη για το πώς μπορούν να συναυθούν και να ενσωματωθούν ε, ε, ε, λογικά τα διασυνοριακές εταιρικέ συμφωνίες στο ευρωπαϊκό εργασιακό πλαίσιο. Δίνω ξανά το λόγο στους προσκεκλημένους. Στον κύριο Χόρν καταρχήν. Για τρία λεφτά να πούμε. Ε, πολύ σύντομα. Εγώ μίλησα για τα θεμελιώδη στοιχεία και ότι θα γίνουν διαφορετικές θα εδραιώσουμε διαφορετικές, ε, ίδιες ρυθμίσεις ε, για αυτές τις διασυνοριακές ε, συμβάσεις είναι σημαντικές ιδέες, όμως, ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι και η εκπροσώπησή τους στις διάφορες χώρες παρόλες τις διαφορετικές ιστορικές συνθήκες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη στα οποία εγκασίστανται οι εταιρείε, θα πρέπει οι εργαζόμενοι πάντοτε να έχουν την ασφάλεια της, ε, των συνθήκων εργασίας. Να ξέρουν δηλαδή ότι εκπροσωπούνται σωστά στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο. Υπάρχουν, ε, όπως είπα, οράματα για μια πλήρη εναρμόνιση, όμως εδώ αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Εγώ θέλω μια δημοκρατική Ευρώπη των πολιτών, των ανθρώπων. Αυτό, σε αυτό συμφωνώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σε εταιρείε και ε, οι εργαζόμενοι, ακόμα και στη Γερμανία βέβαια, αντιμετωπίζουν έναν μεγάλο ανταγωνισμό από την Ισπανία, από τη Γαλλία, από τη Βρετανία. Πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να περιορίσουμε, κάπως να χαλιναγωγήσουμε τους εργοδότες και σε υπερβολικές απαιτήσεις. Και αυτό ακριβώς ε, σε αυτό το σημείο μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο ε, μέσω του, της ενίσχυσης του κοινωνιακού διαλόγου. Τα είπα πολύ γρήγορα. Μπα. Σας ευχαριστώ για τη λακωνικότητά σας. Γιατί από εδώ και πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε αγγλικά, εκτός και αν διερμηνείς μας δώσουν λίγο χρόνο επιπλέον. Ακόμα εδώ είναι. Ε, μιλήστε σε όποια γλώσσα θέλετε, κύριε Ροντρίγκε. Για τρία λεφτά επίση Αγγλικά ή ισπανικά τελικά. Ισπανικά. Για να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο εισηγητής για την ε, ε, ανάγκη να διαθέτουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ε, διασυνοριακές συλλογικές συμβάσεις και για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα που έθεσε ο κύριος Μιούλ. Βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε ορισμού η οπτική μας πρέπει να είναι διασυνοριακή, όχι εναρμόνισης, που δεν είναι εναρμόνιση που κάτι που δεν θα ήταν και εφικτό. Τα διασυνοριακά συστήματα ε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν αλλάζουν, και αλλοιώνουν τα εθνικά συστήματα συλλογικής, συλλογικών συμβάσεων. Βέβαια, ε, υπάρχουν κάποια κοινά θέματα ε, όπως πληρωμένες διακοπές κλπ. που προ, που δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτά μπορούν να τύχουν διαπράγματα σε εθνικό ή κλαδικό επίπεδο. Συνεπώς, ανάγκη δημιουργίας ενός ε, ευρωπαϊκού ε, νομικού ή μη νομικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις. Προφανώς δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπιμότητα, ναι, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο για να αποτρέψουμε ε, συγκρούσεις και διαφορές. Για παράδειγμα, αν οι εργαζόμενοι μιας γαλλικής πολυεθνικής ε, που ε, ε, συνυπογράψουν με τους εργοδότες και τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες μια συμφωνία, αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να γίνει δεκτή από ένα Γάλλο δικαστή. Ε, και, θα, και αν υπάρξει θέμα ερμηνείας αυτής της συμφωνίας θα μπορούσαν ε, να κατατεθούν 200 ή 300 ε, προσφυγές σε γαλλικό δικαστήριο. Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν, δεν είναι θεωρητικό μόνο. Και πρέπει να το αποτρέψουμε. Τέλος, να πω ότι είναι σκόπιμο επειδή η συνθήκη της Λισαβόνας στα άρθρα 152 μέχρι 155 προάγει την ευρωπαϊκή συλλογική διαπραγμάτευση. Θα πρέπει βέβαια αυτή να γίνεται θίγοντας ώστε να το λιγότερο το, τις εθνικές διαπραγματεύσεις και υπάρχουν προτάσεις για να γίνει κάτι τέτοιο έτσι ώστε οι διασυνοριακές συλλογικές συμβάσεις να έχουν εθνικές επιπτώσεις υπάρχουν προτάσεις με ισχυρά επιχειρήματα προτάσεις για ενοποίηση της νομοθεσίας ή πολύ πιο απλές ε, και ήπιες που δεν δημιουργούν προβλήματα. Συνεπώς, ε, ας μην ξεκινήσουμε ε, από τη στέγη, την κατασκευή του σπιτιού, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα θεμέλια, να δούμε ποια προβλήματα θέλουμε να λύσουμε και μετά να προχωρήσουμε στο σύστημα. Ευχαριστώ.